να ξεκινήσουμε με το σημείο 14 της Μεσής Διατάξεως προς μια παρουσίαση μελέτης αναφορικά με τις ε, επιστροφές ιδιοκτησίας. Το πρώτο θέμα που θα εξετάσουμε είναι αυτό της ε, ιδιωτικής ε, περιουσίας τα ακίνητα για την Βοσνία Ριζαγοβίνη θα δώσω το λόγο στην κυρία Μικαέλα Σάλομον και τον, στον Τόμις Μπόρις οι οποίοι θα μας μιλήσουν για το ίδιο θέμα. Θα ήθελα να σας ζητήσω να τηρήσετε τον χρόνο ομιλίας για κάθε έκθεση. Έχουμε προβλέψει 15 λεπτά. Επειδή υπάρχουν δύο παρεμβάσεις αναπαρουσίαση, θα επιμηκύνουμε ε, τον χρόνο 20 λεπτά λοιπόν για κάθε παρουσίαση και παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο. Yeah, does it work? Fine. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie... Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι να αρχίσω, θα αρχίσω εγώ την παρουσίαση. Σκεφτήκαμε στην παρουσίαση πρώτα να κάνουμε μια ε, ανασκόπηση των βασικών στοιχείων που οδήγησε σε απαλωτριώσεις μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδιαίτερα μετά την ανεξαρτησία ε, ορισμένων βαλκανικών χωρών στα Δυτικά Βαλκάνια. Θυμηθείτε τις συνέπειες ε, του Δευτέρου Παγκοσμίου. Διαπιστώνουμε ότι η κοινωνικοποίηση όλων των παραγωγικών αγαθών αποτέλεσε τον πυρήνα του σοσιαλιστικού οικονομικού μοντέλου. Το οποίο σοσιαλιστικό οικονομικό μοντέλο με πρώτη ματιά φαίνεται να παρουσιάζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες και ε, ε, χαρακτηρίζεται ως κοινωνικό αγαθό σε όλες τις χώρες. Το περιεχόμενο όμως της έννοιας αυτής της έννοιας του κοινωνικού αγαθού διαφοροποιεί το στις επιμέρους χώρες και είχε διαμορφωθεί με διαφορετικό τρόπο. Εδώ έχουμε ιδιαίτερα υπόψη τις χώρες που έχουμε καταπιαστεί η κυρία Σόλομον και εγώ, Νία Ερζεγοβίνη, Κροατία και Κωσυφοπέδιο. Αυτές οι τρεις χώρες ανήκαν στην πρώην Ιουγκοσλαβία το κράτος της Ιουγκοσλαβίας είχε ακολουθήσει άλλη εξέλιξη μετά το 1945 και πιο συγκεκριμένα μετά την ρήξη με το Στάλιν από ό,τι άλλες χώρες. Ιδιαίτερα στα πλαίσια αυτής της μελέτης η Βουλγαρία, Ρουμανία και η Αλβανία. Η διαφοροποιημένη διαμόρφωση λοιπόν του οικονομικού μοντέλου στηρίχθηκε σε διαφορετική αντίληψη της κοινωνικής ιδιοκτησίας, η οποία διαμορφώθηκε ως εξής. Με τον πλέον διαφορετικό τρόπο, ε, λάθος, ε, όχι, δεν, μίλησε, δεν ήθελα να πω για επιστροφή, ήθελα να πω για αφαίρεση της ατομικής ιδιοκτησίας, απαλωτρίωση. Να σημειώσω ότι ιδιαίτερα στην πρώην Ιουγκοσλαβία πάντα και την εποχή μετά το 1945 και μέχρι το 1990 πάντα υπήρχε ατομική ιδιοκτησία και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με άλλες χώρες ε, που έχουμε μελετήσει όπως η Αλβανία όπου ατομική ιδιοκτησία δεν υπήρχε πια καθόλου. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε εδώ με ένα διαδικό σύστημα, ιδιικό σύστημα που υπήρχε στο οικονομικό μοντέλο. Η κοινωνική ιδιοκτησία, το βασικό μοντέλο και Παράλληλα συνυπήρχε και ατομική ιδιοκτησία. Αυτή η κοινωνική ιδιοκτησία θεμελιώθηκε στις απαλωτριώσεις των περιουσιών. Ο Κροάτης νομοθέτης, για παράδειγμα, στη δεκαετία του 90 διαπιστώνει πάνω από 30 διαφορετικά κους τρόπους απαλωτρίασης περιουσιών. Και δεν ε, είναι εξαντλητικό ο κατάλογος, οι 30 είναι οι βασικοί τρόποι απαλωτρίωσης ε, περιουσιών. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι τότε πολιτικοί ηγέτες, η πολιτική εξουσία ήταν πολύ εφάνταστη σχετικά με το πώς θα μπορούσε να απαλωτριώσει τις περιουσίες. Πιο δύσκολο βέβαια είναι έτσι να δούμε με ποιο τρόπο η απολωτριωθήσα περιουσία μετά το 1990 και την ε, αλλαγή θα, μπορούσαν, θα μπορούσε η περιουσία αυτή να επιστραφεί. Και θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη άλλες προϋποθέσεις πλαίσιο όταν μιλάμε για τον τρόπο της επιστροφής των περιουσιών. Μεγάλο ρόλο παίζει εδώ το πώς καταχωριζόταν η περιουσία, τα κίνητα, σε ποιο μητρό καταχωρίζονταν. Στην πρώην Ιουγκοσλαβία έχουμε μια ιδιαιτερότητα που χαρακτηρίζεται από το ότι η χώρα αυτή από πολύ νωρίς ήδη είχε υιοθετήσει ένα μοντέλο που υπήρχε στην Αυστρία και την Ουγγαρία. Στην Αυστρία κυρίως. Ένα μοντέλο που στηριζόταν σε δύο θεσμικούς φορείς, σε δύο, υπήρχε το ε, κτηματολόγιο και ο, βασικός κατάλογος με διαφορετικές λειτουργίες. Το, ο βασικός κατάλογος ήταν και είναι ε, η καταχώρηση η οποία είναι σημαντική για την νομική κυριότητα της περιουσίας, ενώ το κτηματολόγιο για τα πρακτικά δεδομένα ενός ακινήτου. Και στην πρώην Ιουγκοσλαβία αυτό ίσχυε σε όλες τις επιμέρους δημοκρατίες. Ήδη από το 1931 ε, ίσχυε το σύστημα αυτό. Παντού. Μία εξαίρεση ήταν de facto το κοσυφοπαίδιο, γιατί το Κόσοβο μετόχια τότε, εκεί ίσχυε το παλιό σύστημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που ήταν, ε, στηριζόταν σε διαφορετικό τρόπο καταχώρησης. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Σας τα λέω γιατί όλα τα μέτρα απαλωτρίωσης των περιουσιών μετά το 1945 στην πρώην Ιουγκοσλαβία καταχωριζόταν στο βασικό κατάλογο. Οπότε, εάν δούμε τον κατάλογο αυτό, γνωρίζουμε πολύ καλά πάνω σε ποια βάση έγινε η απαλωτρίωση της περιουσίας. Έτσι, μας διευκολύνει αυτό να καθορίσουμε και τον τρόπο της επιστροφής πλέον της συγκεκριμένης περιουσίας. Το λέω αυτό γιατί και για τα δύο μέρη αυτής της μελέτης έχει σημασία και για το κομμάτι που αφορά την περιφερειακή σύγκρουση, η διένεξη, αλλά και το κομμάτι εκείνο το οποίο θίγεται από την ε, πολιτική αλλαγή και μόνο. Το ζήτημα της επιστροφής γενικά από νομική άποψη, και εγώ είμαι νομικός, Είναι λοιπόν το θέμα της επιστροφής ένα θέμα το οποίο πρέπει να, βεβαίως πρέπει να λυθεί σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά σε πολιτικό επίπεδο δεν είναι πολύ δύσκολο το ζήτημα, γιατί σε τελευταία ανάλυση μπορεί κανείς να ταχθεί υπέρ δύο συστημάτων. Είτε θα λάβει χώρα η επιστροφή πριν από την αποζημίωση ή θα μπορεί ο νομοθέτης να πει θα γίνει αποζημίωση και κατ' εξαίρεση μόνο θα προβλέπεται η δυνατότητα επιστροφής του ιδίου του ακινήτου της περιουσίας. Αυτές οι δύο προσεγγίσεις είναι κυρίαρχες σε όλες τις χώρες, όχι μόνο σε αυτές που εξετάζουμε σήμερα, αλλά σε όλες τις χώρες που προέκυψαν από το πρώην κομμουνιστικό σύστημα της οικονομίας. κατά την επίλυση του θέματος της επιστροφής και πώς μπορεί αυτή να λάβει χώρα. Οι, Βοσ... οι τρεις χώρες που εξετάσαμε, Βοσνία, Τζεγοβίνη, Κωσυφοπέδιο και Κροατία, πάνω στη βάση, ε, ε, λόγω του πολέμου, ακολουθήθηκαν διαφορετικές διαδικασίες και εξελίξεις. Οι διαφορετικές αυτές εξελίξεις αποτελούν και το πυρηνικό πρόβλημα ε, απέναντι στην υιοθέτηση μιας ενίας προσέγγισης. Γιατί? Γιατί η Κροατία ακολούθησε ένα δρόμο που από... είναι... Ε, πολύ συστηματικός νομικός, δηλαδή προσπάθησε το θέμα της επιστροφής να το λύσει από κοινού, μαζί με το πώς καταρχήν καταχωρίζονται τα ακίνητα, συνέδεσε τα δύο θέματα και συνέδεσε επίσης και ένα άλλο θέμα, δηλαδή πώς εμπράγματες αξίες, τα property rights, αυτές οι εμπράγματες αξίες πώς διαμορφώνονται και τα δικαιώματα επί εμπραγμάτων αξιών, πώς μπορούν να διαμορφωθούν επαρκώς. Τα τρία αυτά στοιχεία συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους. Δεν μπορεί δηλαδή να δούμε μόνο τα δικαιώματα επιστροφής, θα πρέπει να τα βλέπουμε πάντα πάνω στη βάση της καταχώρησης των ακινήτων και το πώς γενικά ρυθμίζονται θέματα εμπράγματων αξιών. Η Κροατία είναι η μόνη χώρα η οποία επέλεξε αυτήν την ενιαία προσέγγιση η οποία ταυτόχρονα τον Ιανουάριο του 1996 τα ρύθμισε και τα τρία. Στη Βοσνία ήταν πιο, δύσκολα τα πράγματα λόγω του πολέμου, της πολεμικής αντιπαράθεσης που διήρκεσε πολύ περισσότερο. Και στο το Κωσυφοπαίδιο βεβαίως που εκεί ε, αντιμετώπισε πόλεμο. Ούτε όμως η Βοσνία, ούτε το Κωσυφοπαίδιο μέχρι τώρα δεν κατάφερε να ε, επιλέξει την ε, κροατική προσέγγιση. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ακόμα υποφέρει γιατί δεν μπορεί να βρει ποιο είναι υπεύθυνο για θέματα ρύθμιση εμπράγματων αξιών. Δεν υπάρχει σαφής απάντηση. Ποιοι θα είναι. Θα είναι το ομοσπονδιακό κράτος ή τα entities ή άλλοι φορείς. Ε, αυτό το θέμα ακόμα δεν έχει ε, επιληθεί και κατά τις συζητήσεις ε, για το εμπράγματο δίκαιο αυτά τα θέματα δημιούργησαν αντιπαραθέσεις. Στο δέκο ψηφοπαίδιο υπάρχουν προβλήματα λόγω το, της μεγάλης κλίμακας εκτοπισμού το 98-99 το νεαρό κράτος μετά το 2008 δεν είχε ακόμα τη δυνατότητα να προβεί σε νέες ρυθμίσεις Τώρα ε, προχωρούν σε ένα σχέδιο του δικαίου. Γενικά, και θα κλείσω τις παρατηρήσεις μου, γενικά τι ε, θα, μπορούσε κανείς να συστήσει στα θέματα αυτά. Η πρώτη σύσταση, η συμβουλή, είναι να μην χωριστά το θέμα της επιστροφής χωρίς να συμπεριληφθεί το θέμα της καταχώρησης των ακινήτων και το θέμα του εμπράγματου δικαίου. Αυτή είναι μια πρώτη σημαντική προσέγγιση. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση τι μπορεί να κάνει, δηλαδή ε, και τι να παρέχει, όχι οικονομικά, στο θεσμικό επίπεδο εννοώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δώσει μια συμβολή θεσμική μέσα από τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης και τα σχετικά σύμφωνα αφού θα μπορούσαν εκεί να ληφθούν υπόψη και τα ζητήματα αυτά ούτως ώστε να διευκολυνθεί μια προσέγγιση των χωρών αυτών προς τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί σε τελευταία ανάλυση ο απότερος στόχος όλων αυτών των μέτρων ποιος είναι. Να επιτευχθεί διαφάνεια στο ε, δίκαιο περιουσιών, ούτως ώστε να υπάρχει και νομική ασφάλεια που σήμερα δεν υπάρχει στις τρεις χώρες, ούτε στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, ούτε στο Κωσυφοπαίδιο, ούτε στην Κροατία για διαφορετικούς λόγους σε, κάθε χώρα αλλά και για τις τρεις ισχύει ότι η, ε, το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι οι ανεπάρκειες στη διοίκηση και με, αυτά, με αυτές τις παρατηρήσεις κλείνω την εισαγωγή μου και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και διευκρινήσεις. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην καθηγήτρια Σάλαμον. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω την παρουσίαση με δύο βασικά ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξή. Το διεθνέ δίκαιο προβλέπει το δικαίωμα αποκαταστάσεω ιδιοκτησία για αποζημίωση. Δεύτερο ερώτημα. Ποιο ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και ποιο θα μπορούσε να είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω στη διαδικασία αποζημιώσης και επιστροφή ιδιοκτησίας στην πρώην Ιουγκοσλαβία, στις χώρες που ασχολήθηκε η μελέτη Βοσνία Ζεγοβίνη, Κροατία και Κόσοβο. Όσον αφορά το διεθνές δίκαιο, δύο τομεί του διεθνούς δικαίου ασχολούνται με το θέμα. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει γενική συνένεση κατά πόσο ένα δικαίωμα επιστροφή ιδιοκτησία ή αποζημίωση υπάρχει σαν έννοια. Αλλά ε, αποζημίωση, επιστροφή έχει αποφασιστεί από διάφορους δικαστικούς και δικαστικούς φορείς και από φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό της αποζημίωσης και της επιστροφής ιδιοκτησίας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει επιδικάσει αποζημίωση ή επιστροφή σε περιπτώσεις που αφορούν απολατριώσεις κατά τη διάρκεια κομμουνιστικού καθεστώτος, κατά τη διάρκεια σύγκρουσης ή πολέμου στην πρώην Ιουγκοσλαβία, στη Βόρεια Κύπρο και ε, στην Τουρκία, με βίους εκτοπισμού στην Τουρκία. Άρθρο 1 του πρωτοκόλου 1 της συμβάσεως αναφέρει αυτό το θέμα και το δικαίωμα στη δίκαια δίκη που αναφέρεται στο άρθρο 6 της συμβάσεως. Αυτά τα δικαιώματα, αυτές οι υποθέσεις αφορούσαν κυρίως περιπτώσεις όπου ελήφθη απόφαση, αλλά δεν εκτελέστηκε επί μακρά χρονική περίοδο. Οπότε το άτομο επί για το οποίο είχε επιδικαστεί αποζημίωση και επιστροφή ιδιοκτησίας και δεν μπορούσε τελικά να αποκτήσει την περιουσία του. Άλλος φορέας είναι ο ΙΕ, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το ΙΕ, άλλο φορέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτή η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το ΙΕ, θεώρησε ότι το δικαίωμα στην ισοτιμία στη Διεθνή Σύμβαση για πολιτικά και αστικά δικαιώματα παραβιάστηκε σε διάφορες υποθέσεις σχετικά με τη Τσεχική Δημοκρατία αφορούσε απαλωτριώσει κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και κατά τη διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Τσεχική Δημοκρατία, διότι η τσεχική νομοθεσία έκανε διάκριση μεταξύ αλλοδαπών και ημεδαπών και δεν ήταν δυνατόν οι αλλοδαποί να τύχουν από κατάσταση επιστροφής. Άλλοι φορείς διεθνούς δικαίου, διάφορες επιτροπές που ασχολήθηκαν οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα η Επιτροπή για την καταπολέμηση των ρατσιστικών διακρίσεων και κατά των διακρίσεων κατά των γυναικών, αυτές οι επιτροπές δεν μπορούν να λάβουν δεσμευτικές αποφάσεις. Όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορούν να προβούν σε ανακοινώσεις αν η χώρα έχει επικυρώσει ή έχει δεχτεί αυτή τη δικαιοδοσία και μπορούν να γενικές συστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι είναι λιγότερο αποτελεσματική φορείς από ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το δεύτερο τμήμα τώρα του διεθνούς δικαίου αφορά τις χώρες ξεχωριστά, κατά χώρα. Νόμος κατά χώρα ή που αφορά πρόσφυγες ε, ή εκτοπισμένους. Παραδείγματο χάρη, το δικαίωμα επιστροφής και αποζημιώσεως μπορεί να βρεθεί στη συμφωνία, τη ε, συμφωνία του Dayton στο παράρτημα 7 για τη Βοσνία Ζεγοβίνα και στη συμφωνία την αντίστοιχη για την Κροατία, στο σχέδιο Συμφωνία του Ραμπουγέ δικαίωμα επιστροφής ε, προβλέπεται και έχει αποσημείωση και στο σχέδιο Ατισάρι για το Κωσυφοπαίδιο. Επιπλέον, υπάρχει άλλη διεθνή συμφωνία η οποία ασχολείται με θέματα ιδιοκτησία στην πρώην Ιουγκοσλαβία, η συμφωνία για θέματα διαδοχής κληρονομιάς Παράτημα G λατινικό λέει ότι όλες οι νομικές, νόμιμες μεταφορές υποπίεση μετά την 31η Δεκεμβρίου του 1990 θεωρήθησαν ως ε, κενές περιεχομένου, άκυρες. Αυτή η νευτική συμφωνία αφορούσε την επιστροφή και αποζημίωση ε, και ε, διεκπεραιώθηκε στα πλαίσια του διεθνούς υπείου δικαίου που εμπεριέχεται σε ψηφίσματα της Γενικής Συνελεύσεως του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, παραγματος χάρη, Ψηφίσματα αφορούν κάθε χώρα ξεχωριστά, Βοσνία, ε, Κωσυφοπέδιο, Κροατία και η αρχή Πινέιρο για θέματα στέγασης και επιστροφής ιδιοκτησίας για τους πρόσφυγες και τους εκτοπιστέντες. Οι διεθνείς οργανισμοί όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΑΣΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Πατιαρμοστία για τους πρόσφυγες και διάφοροι άλλοι φορείς ασχολήθηκαν με θέματα επιστροφής περιουσιών μέσω των αρμοδίων φορέων τους, στο δεύτερο τμήμα. Της παρουσιάσεως αυτής που κάνω θέτει ένα θέμα, ένα ερώτημα. Ποιο ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και ποιο θα μπορούσε να είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω όσον αφορά την επιστροφή των ιδιοκτησιών και τη διαδικασία αποζημιώσεων για αυτό το ερώτημα γίνεται μια βασική διάκριση. Πρέπει να γίνει μια βασική διάκριση μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ κρατών που έχουν συμφωνία συνδέσεω, όπως είναι η Κροατία τώρα, συμφωνία σύνδεση με τη Βοσνία δεν έχει τεθεί σε ισχύ ακόμα και τρίτο χώρε χωρί συμφωνία σύνδεση, όπως είναι το Κωσυφοπέδιο, το Κόσοβο. Γιατί γίνεται αυτή η διάκριση, γιατί είναι αναγκαία αυτή η διάκριση, διότι διάφορες πηγές ευρωπαϊκού δικαίου, ευρω... δικαίου της Ευρωπαϊκής εφαρμόζονται σε αυτές τις χώρες. Για ε, τα κάτι μέλη ε, ισχύει ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ενώσης εκτός από αυτοεξαιρέσεις κρατών. Όπως διάφορες αυτοεξαιρέσεις opt-out από τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που περιέχεται στις συνθήκες της Αβώνας. Μετά, Υπάρχουν και χώρες με συμφωνία σταθερότητας. Εφαρμόζεται έμεσα το δίκαιο της Ευρωπαϊκή Ενώσεως μέχρι νομικών υποχρεώσεων για την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου. Όσον αφορά τα κράτη-μέλη, η διανομή των εξουσιών μεταξύ ενώσεως και κρατών μελών βασίζεται, όπως όλοι γνωρίζετε, επί της αρχής της εκχωρηθήσης εξουσίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυτές τις αρμοδιότητες μόνο, οι οποίες τις ανατίθενται ρητά από τα κράτη-μέλη μέσω συνθήκων, ε, διεθνών συνθήκων. Όμως, αυτή η αρχή έχει διαβρωθεί κατά κάποιο τρόπο σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που εφάρμοσε την αρχή των υπονοουμένων αρχών ε, και μια άλλη αρχή ε, ποια είναι η πιο αποτελεσματική απόφαση. Και έτσι διευρύνθηκε στην πράξη η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν υπάρχει διάταξη που ρητά δίνει την αρμοδιότητα για θέματα διοκτησίας στην κοινότητα. Αντιθέτως μάλιστα υπάρχει το άρθρο 345 που αναφέρει ότι η συνθήκη δεν εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των κρατών μελών πως εφαρμόζουν την αρχή της ιδιοκτησίας. Αυτό σημαίνει αρνητική αρμοδιότητα για την Ένωση. Αυτό επιχειρηματολογήθηκε από κάποιους ειδικού για τα νομικά θέματα, εξαρτάται, διότι το σύστημα της ιδιοκτησίας δεν είναι πολύ σαφές, δεν είναι καλά καθορισμένο. Ίσως μπορεί να ερμηνευθεί πάρα πολύ γενικά, να καλύπτει ιδιοκτησία και όλα τα συναφή δικαιώματα ίσως να ερμηνευτεί πάρα πολύ στενά, να καλύπτει μόνο το κατά πόσο ένα, μια ιδιοκτησία ανήκει σε ιδιώτη ή στο κράτος, μπορεί να κρατικοποιηθεί ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, ο εθνικό νομοθέτη θα πρέπει να εφαρμόσει τι βασικέ αρχέ τη συνθήκη, την απαγόρευση της διάκριση λόγω εθνικότητα, τι βασικέ ελευθερίε και του νόμου περί ανταγωνισμού. Από την άλλη πλευρά τώρα, ο κοινοτικό νομοθέτη μπορεί να περιορίσει την ιδιοκτησία, την ιδιωτική, για να πετύχει σημαντικού κοινοτικού στόχου. Ποιοι είναι οι κοινοτικοί στόχοι που είναι σημαντικοί, ποιοι θα μπορούσαν να είναι αυτοί οι σημαντικοί κοινοτικοί στόχοι, παραδείγματο χάρη. Ο στόχο να επιτευχθεί πολύ ε, ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, άρθρο 3 της συνθήκης. Δηλαδή, μπορεί να πει κανείς, επιχειρηματολογώντας, ότι η κοινότητα μπορεί να παρέμβει σε εθνική νομοθεσία για να ρυθμίσει την αγορά γεών, ούτως ώστε να πετύχει την ασφάλεια της αγοράς και την ασφάλεια της ιδιοκτησίας. Μόνο έτσι μπορεί η αγορά γεών να λειτουργεί σωστά, κτήματα αγορά, και μόνο αν λειτουργεί κτήματα αγορά θα μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος μιας οικονομίας αγοράς με κοινωνικό πρόσωπο είναι ένα θέμα ερμηνείας με άλλα λόγια και κατά πόσο υιοθετεί κανείς μια ευρεία ή μη ευρεία ερμηνεία. Διότι το θέμα αυτό, η έννοια της ιδιοκτησίας είναι αρκετά ασαφής. Όπως προανέφερα, οι θεμελιώδεις ελευθερίες εμπεριέχουν το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, η κάθε μία της ελευθερίας. Πέραν αυτού, επιπλέον, η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που είναι νομικά δεσμευτική, από όταν ετέθη σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας, εμπεριέχει δικαιώματα για διεκτησία ισοτιμία, μη διάκριση, για δίκαιη δίκη και για γεωθωτικά μέτρα, αποζημιώσεις τα περισσότερα δικαιώματα, αυτά που προβλέπονται, έχουν το ίδιο περιεχόμενο, το ίδιο περιεχόμενο όπως στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αυτό αναφέρεται στις, στις επεξηγήσεις της χάρτας. Όσον αφορά το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, παραδείγματος χάρη, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη την αρχή της νόμιμης προσδοκίας. Δηλαδή να πιστεύει ο πολίτης στη συνέχεια των νομικών θέσεων που θεσπίζονται από τον νομοθέτη αν η ιδιοκτησία δεν είναι ασφαλής, δεν είναι σίγουρη σε μια χώρα. Γιατί, διότι η χώρα το χάρη ε, δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία επιστροφών τη μετακομμουνιστική. Μπορεί κάποιος να αξιώνει δικαιώματα για ε, ιδιοκτησία και να κρεμούν αυτά. Εκεί δεν υπάρχουν νόμιμες προσδοκίες όσον αφορά μια συγκεκριμένη γη, σε αυτή την περίπτωση που αναφέρω. Θα έρθω τώρα στη βασική σύσταση, στις βασικές συστάσεις όσον αφορά το διεθνές δίκαιο και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Βεβαίως η αμοιβαιότητα, η αρισιμότητα θα πρέπει να εξακολουθεί να ισχύει μέσω των μέσων του Συμφώνου Σταθερότητας και Σύνδεσης και είπατε εκπρόσωπο στη Βοσνία πρέπει να ασκεί τις εξουσίες και οι εξουσίες της Γιούλεξ στο Κωσυφοπέδιο έχει δυνατότητες παρέμβασης που προσωμιάζουν με εκείνες του του εκπροσώπου συνεχής βοήθεια από πλευράς Ευρωπαϊκή Ενώσεω είναι σημαντική οικονομική βοήθεια, κυρίω για δημιουργία δυναμικού και καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς και να σχεδιάζει μηχανισμούς επιβολής του νόμου και να κάνει αποτελεσματική την επιβολή και εφαρμογή του νόμου, κάποιες δυνατότητες εφαρμογής πολιτικής να υποστηρίζονται, όπως επιστροφή ε, πριν αποζημίωση να λαμβάνει κανείς σοβαρά υπόψη, να διορθώνει, να αποκαθιστά, να βοηθά ε, δευτερεύοντες, ε, διαμένοντες με διάφορες αξιώσεις που έχουν και μετά τη δυνατότητα να αξιώσει κανείς επιστροφή στους κληρονόμους, μη πολίτες και μη μονίμους κατοίκους, όποτε αυτό προβλέπεται από την νομοθεσία. Επιπλέον, σε κάποιες χώρες, ίσως να χρειαστεί να υπάρχουν συστήματα που παρέχουν πληροφορίες για τα εδάφη με διάφορα επίπεδα ιδιοκτητών και διάφορες αξιώσεις. Ας πούμε, οι ιδιοκτήτες πρώτου κομμουνιστικού καθεστώτος θα πρέπει να φαίνονται στο σύστημα αυτό και κρεμούσε αξιώσεις για κάποιες ιδιοκτησίες θα πρέπει και αυτές να φαίνονται, οπότε η ιδιοκτησία θα γίνεται πιο διαφανής. Αυτό το σύστημα θα πρέπει να είναι προσβάσιμο, η προσβασιμότητα είναι σημαντική. Κάτι παρόμοιο ξεκίνησε με το Ευρωπαϊκό Σύστημα για την Υπηρεσία για τις ΓΕΕΣ. Μόνο μερικές χώρες συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το κτηματολόγιο και από ό,τι γνωρίζω αντίθετα σε αξιώσεις για συγκεκριμένη ιδιοκτησία ε, δεν αποφασίζονται, δεν ρυθμίζονται εκεί και θα πρέπει να υπάρχει και μια βάση δεδομένων με νομικές πληροφορίες. Αυτό είναι σημαντικό και εδώ κλείνω την παρουσίασή μου και ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα περάσουμε στη δεύτερη μελέτη και να δώσω το λόγο στην κυρία Λάουδα Στέφαν. Η δεύτερη μελέτη πάνε σε ζητήματα ιδιοκτησίας αφορά την αλλαγή καθεστώτος στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Thank you very Ευχαριστώ πολύ. Αυτή η μελέτη εξετάζει την ατομική ιδιοκτησία μετά την αλλαγή, την πολιτική, μετά το πέρασμα του σοσιαλιστικού ή κομμουνιστικού καθεστώτος στην σημερινή κοινωνία και το σύστημα. Οι χώρες που καλύπτονται από τη μελέτη είναι πιο πολύ άριθμες από ό,τι στην προηγούμενη μελέτη. Κοιτάμε Αλβανία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Ρουμανία και Σερβία. Βλέπετε ότι οι χώρες είναι σε διαφορετικά στάδια ή φάσεις σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιες είναι ήδη ε, κράτη-μέλη, Βουλγαρία, Ρουμανία, άλλε είναι υποψήφιε, άλλε είναι δυνητικά υποψήφιες. Η δομή τη μελέτη έχει ω εξή. Καταρχήν κάνουμε μία σύνοψη, μετά μία εισαγωγή. Μετά έχουμε το πρώτο τμήμα που εξετάζει το Διεθνές Δίκαιο και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη δική μας περίπτωση το Διεθνές Δίκαιο σημαίνει Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γιατί στην περίπτωση αλλαγής καθεστώτων έχουμε λιγότερες διεθνείς ρυθμίσεις σε σχέση με την μετασυγκρουσιακή ε, περίοδο μεταξύ κράτους και προσφύγων. Δεύτερο μέρος, ανάλυση της επιστροφής περιουσιών στις έξι χώρες. Η ανάλυση ακολουθεί την ίδια δομή περίπου με τις έξι χώρες, με μια ανασκόπηση μετά θέματα ε, εθνικοποιήσεων ή αποθηνικοποιήσεων επιστροφών, τι έγινε με την επιστροφή μετά την αλλαγή, ήδη επιστροφή ανάλογα με το είδος της, του περιουσιακού στοιχείου. Σε πολλές χώρες η επιστροφή αγροτικών γεών ή αστικών περιοχών είναι χωριστά. Σε ορισμένες χώρες υπάρχουν διαφορές μεταξύ επιστροφής γεών και επιστροφής κτηρίων και κάθε μελέτη περίπτωσης ε, συνοδεύεται από σειρά συμπερασμάτων για τις χώρες, για κάθε χώρα. Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τι μας ενδιαφέρει ως επιτοπλίστων εδώ. Το άρθρο 1, πρωτόκολλο, πρωτόκολλο 1 που μιλάει για δικαιώματα περιουσιών και το άρθρο 6 το οποίο καλύπτει την δίκαιη δίκη. Εδώ έχουμε καταγράψει τα είδη των ε, προσφύγων στο δικαστήριο και αξιώσεων από όλες τις χώρες που καλύπτει η μελέτη. Μιλάμε για μία επιβολή των τελεσίδικων αποφάσεων. Μιλάμε επίσης ε, για περιουσία που αφαιρέθηκε ενώ υπήρχε προστασία του μισθωτή. Μιλάμε επίσης για δικαστήρια ως επιτοπλίστων τα ανώτατα τα οποία ε, αναιρούν άλλες αποφάσεις των δικαστηρίων, αποτυχία της διοίκησης ε, να αποζημιώσει σύμφωνα με τους ε, κανόνες και εθνικούς νόμους και πρόσβαση στα δικαστήρια προκειμένου περί επιστροφής κατασχεμένης περιουσία είτε λόγω υψηλών ταπανών ή άλλων εμποδίων. Πρέπει να πούμε ευθύ εξ αρχή ε, ότι η αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καλύπτει ό,τι συμβαίνει αφού υπογράψει τη σύμβαση η χώρα. Την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εννοώ. Και έχουμε καταγράψει στη μελέτη τα έτη ε, κατά τα οποία συνέβη αυτό, δηλαδή η προσχώρηση στη σύμβαση για, από κάθε χώρα. Κάποια στατιστικά στοιχεία εδώ που εξετάζουν την κάθε χώρα χωριστά, αριθμό ε, ετήσεων που εκκρεμούσαν στο τέλος του 2009, έπρεπε να έχουμε αυτό το έτος αναφοράς το 2009 γιατί τότε είχαμε, από εκεί μόνο είχαμε διαθέσιμα δεδομένα όταν τελειώσαμε τη μελέτη. Είδαμε πόσες αιτήσει λοιπόν θεωρήθηκαν απαράδεκτες, αριθμός των αποφάσεων του δικαστηρίου, πόσες παραβιάσεις διαπιστώθηκαν βάσει του άρθρου 1 πρωτόκολλο 1 και αν σε σχέση με τις χώρες θεώρησε το δικαστήριο ότι υπάρχει συστημικό πρόβλημα με το ζήτημα της επιστροφής των περιουσιών. Για την Αλβανία, Βοσνία, Ρουμανία ε, εντοπίστηκε πρόβλημα συστημικό από το δικαστήριο. Τώρα θα μιλήσουμε ε, για τις ιδιαιτερότητες των χωρών όταν περάσουμε στις μελέτες των περιπτώσεων. Εδώ να πω μόνο ότι για τη Σερβία το γεγονός ότι το δικαστήριο δεν διαπίστωσε συστημικό πρόβλημα ακόμα δεν σημαίνει και τίποτε γιατί η Σερβία δεν άρχισε καθόλου να επιστρέφει περιουσίες. Οπότε τι να βρει το δικαστήριο, τι συστημικό πρόβλημα να βρει. Δεν θα υπησέλθω σε λεπτομέρειες σχετικά με τις αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτό το ανέφεραν στην προηγούμενη μελέτη οι συνάδελφοι. Θα ήθελα όμως να αναφέρω ένα φορέα που είναι καλός, είναι ο φορέας θεμελιωδών δικαιωμάτων, που διεξάγει έρευνες και διαμορφώνει άποψη και γνωμοδοτεί για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι το θέμα των δικαιωμάτων επιπεριουσιών ή του δικαίου ιδιοκτησίας μπορεί να καλυφθεί επαρκώς από το φορέα αυτόν. Τώρα, ας πάμε στις χώρες. Εδώ ένας κατάλογος θεμάτων που θεωρούμε ότι ισχύουν λίγος πολύ στις χώρες που εξετάσαμε. Το πρώτο μείζον θέμα είναι η καθυστερημένη έγκριση πολιτικών επιστροφών περιουσιών. Να αναφέρω εδώ ότι η καθυστέρηση δεν αναφέρεται σε κάθε είδους ιδιοκτησία, γιατί αυτό που είδαμε είναι ότι όσο λιγότερες είναι οι διαφορές και αντιπαραθέσεις ε, επιπεριουσιακών, τόσο πιο πιθανό ήταν να ρυθμιστεί το ζήτημα της επιστροφής στην αρχή της δεκαετίας του 90, όπως με τις γεωργικές γέες. Η επιστροφή γεωργικών γεών έγινε ευκολότερα και στην αρχή της δεκαετίας του 90, ενώ καθώς προχωρούμε και πάμε σε επιστροφή αστικών ε, κτηρίων, σε μεγάλες πόλεις κλπ, εκεί περιπλέκονται περισσότερο τα πράγματα ασαφής και απρόβλεπτη πολιτική επιστροφών. Είδαμε μετατοπίσεις στις πολιτικές επιστροφής περιουσιών, μετατοπίσεις που ε, δυσκόλεψαν πάρα πολύ την διοίκηση, γιατί αν η πολιτική αλλάζει κάθε τέσσερα χρόνια, είναι πάρα πολύ δύσκολο η διοίκηση να παρακολουθεί τις αλλαγές και έχουμε θέματα εφαρμογής του νόμου και χρονικές καθυστερήσεις. Επίσης, αδύναμη ε, θεσμική ικανότητα της διοίκησης. Αυτό είναι οριζόντιο θέμα, δεν αφορά μόνο τις επιστροφές περιουσιών, αλλά τις επηρεάζει. Γιατί ζητάμε από τη διοίκηση να αναλάβει το καθήκον αυτό, ενώ η διοίκηση έχει τα δικά της βάσανα και ελλείψεις. Συστημικά προβλήματα στη δικαστική εξουσία επηρεάζει επίσης την επιστροφή. Λόγω των απρόβλεπτων πολιτικών και των συχνών αλλαγών πολιτικών βλέπουμε ε, επικαλυπτόμενα δικαιώματα επί του ιδίου ακινήτου. Αυτό συμβαίνει συχνά σε ορισμένες χώρες. Τέλος το θέμα της αποζημίωσης που θεωρούμε ότι είναι αναποτελεσματική ως ένα βαθμό. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση τι μπορεί να κάνει. Όπως είπα στην αρχή, οι χώρες δεν είναι οι ίδιες όλες και βρίσκονται σε διαφορετική χρονική στιγμή στη σχέση τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε είναι και διαφορετικό το τι μπορεί να κάνει η Ένωση στις χώρες, σε κάθε χώρα. Να συνεχίσω με τη χρήση του παραδοσιακού μηχανισμού παρακολούθησης και των συστημάτων των όρων που τίθενται. Πρέπει επίσης να δούμε πάλι την νομοθεσία και την εφαρμογή της νομοθεσίας, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές ε, βλέπουμε σε χώρες να υπάρχει νομοθεσία αλλά δεν εφαρμόζεται. Επίσης, ε, να ζητήσουμε από τις ε, κυβερνήσεις προγράμματα δράσης, συγκριτικές αξιολογήσεις, κατανομή κονδυλίων του προϋπολογισμού, υπεύθυνους θέσμου. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να δούμε το κόστος. Ιδιαίτερα στη σημερινή ε, κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν να διερευνήσουμε μηχανισμό χρηματοδότηση. Αυτό θα πρέπει να είναι αντικείμενο συζήτηση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρών για να δούμε πώ μπορούμε να δούμε θέματα ιδιωτικοποίηση, αμοιβαία κεφάλαια, ε, ειδικά δάνεια με ειδικού όρου, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα ε, τι επιπτώσει που θα έχει αυτό στο δημοσιονομικό έλλειμμα το οποίο, όπως είπα, σε καιρούς όπως η σημερινή είναι ένα θέμα καυτό Τώρα πάμε στις μελέτες των περιπτώσεων των χωρών. Προσπαθούμε με πολύ συμπιεσμένο τρόπο να παρουσιάσουμε τα ευρήματά μας από κάθε χώρα, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ακολουθήσουν και ερωταπαντήσεις, όπου θα σας δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τις αναλυθήσεις χώρες. Στην Αλβανία φαίνεται ότι το 1991-1992 είχαμε τους πρώτους νόμους για την ιδιωτικοποίηση και ε, ως ένα βαθμό υπήρξε ε, μεταφοβίβαση κτηρίων και ε, διαμερισμάτων και αγροτικών γεών. Το 1993 ο πρώτος νόμος για την ε, επιστροφή και την αποζημίωση πρώην ιδιοκτητών, αστικών ακινήτων και το 2000 και Εκεί άρχισαν οι πρώτες επιστροφές. Κοιτάζοντας όμως την επιστροφή βλέπουμε ότι σε επιχειρησιακό επίπεδο λείπουν οι κανόνες, οι κανονισμοί και είναι πολύ δύσκολο η χώρα να προχωρήσει στην πράξη και να προβεί στις επιστροφές. Βοσνία Ερζαγοβίνη. Το 1996 πέρασαν δύο νόμοι στην ε, Σερβική Δημοκρατία για την επιστροφή των περιουσιών και το 1997 ένας νόμος για τις πωλήσει διαμερισμάτων που ε, ε, ήταν κατοικημένα στην ε, Βοσνία Ερζεγοβίνη και στην Σερβική Δημοκρατία. Το 2000 πέρασε νέος νόμος από τη Σερβική Δημοκρατία για τις επιστροφές που αμέσως ακυρώθηκε από το γραφείο του υπάτου εκπροσώπου. Είχαμε δύο νόμους λοιπόν για την επιστροφή και μετά ο νόμος αυτός τέθηκε σε αναστολή. Υπάρχει τώρα ένα νέο σχέδιο που αναλύουμε στη μελέτη και το οποίο εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2009, ένα νομοσχέδιο το οποίο μιλάει για ε, επιστροφή σε είδος και αποζημίωση. Αυτό εξετάζομαι στη μελέτη. Αυτά τα δύο στις χώρες ε, είναι τα δύο συστήματα που συμβαδίζουν. Το πρώτο είναι η επιστροφή σε είδος και μετά η αποζημίωση και μετά καλύπτουν τι κατηγορίε τα είδη περιουσιών που βλέπετε και στη διαφάνεια. Ακόμα δεν έχει εγκριθεί όμω, δεν έχει περάσει το νομοσχέδιο, οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Για τη Βουλγαρία κάνουμε διαφοροποίηση μεταξύ γεωργικών λεών και, γεών και αστικών. Το 1991 ο, εγκρίθηκε ο νόμος για τις περιουσίες και τη χρήση γεωργικών γεών. Μιλάει για επιστροφή σε είδος και αποζημίωση. Το 1992 έλαβαν χώρα τροπολογίες υπέρ της επιστροφής σε είδος και το 1999 τροπολογίες για ε, κάποια ομόλογα αποζημίωσης, ε, κάποια ομόλογα που ελάμβαναν οι δικαιούχοι. Ήταν ξεκάθαρη όμως η διοικητική διαδικασία, οπότε μέχρι το, στο τέλος του 2000 το 99 περίπου τις 100 των γεών είχαν επιστραφεί. Πρέπει να αναφέρουμε όμως εδώ ότι δεν επεστράφησαν όλες οι γέες που είχαν ε, ετηθεί, αλλά δόθηκαν τα ο μέγιστο, δόθηκε ο επιστράφει ο μέγιστος αριθμός οικοπαίδων που πρόβλεπε ο νόμος. Γιατί η Βουλγαρία το 1992 εγκρίθηκε ο νόμος για τις επιστροφές εθνικοποιημένης ε, ακίνητης περιουσίας, ε, με την προϋπόθεση ότι θα εξακολουθούσε να υπάρχει το ακίνητο, η περιουσία, ότι θα ήταν ο ιδιοκτήτης στο κράτος και ότι δεν θα ε, είχε καταβληθεί αποζημίωση όταν είχε γίνει η εθνικοποίηση. Και το 95% μέχρι το 2000 είχε επιστραφεί. Το θέμα των αποζημιώσεων. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ότι υπάρχουν διάφορα είδη αποζημιώσεων. Το πρώτο είναι να ε, δώσει μερίδια σε, εξουσία, ε, διοκτησίες ή μερίδια σε μετοχές επιχειρήσεις ή κάποιες ομολογίες. Ορισμένες μπόρεσαν να ε, παίξουν στο χρηματιστήριο, άλλες ήταν σημαντικές για τη στέγη, άλλες ομολογίες. δόθηκαν ε, για δασικές περιοχές. Πάντως ε, επηρεάζεται το, η αξία των ομολογιών αυτών για αποζημίωση αντισταθμιστικών ομολογιών ε, ανάλογα με τη χρήση τους επηρεάστηκε λοιπόν ε, η αξία των ομολογιών αυτών. Στην Κροατία το 1996 είχαμε τον πρώτο νόμο για την αποζημίωση ε, απαλωτριωμένων περιουσιών από το κομμουνιστικό καθεστώς. Ε, φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούσαν να πάρουν επιστροφή. 71% των απαιτήσεων οριστικοποιήθηκαν και 69% ε, των αιτήσεων αξιώσεων εγκρίθηκαν από τη διοίκηση. Τα προβλήματα που είδαμε είχαν σχέση με εγγενή συγκρούση συμφερόντων μεταξύ αυτών που επρόκειτο να επιστρέψουν τις περιουσίες και που ήταν εκείνοι που ήταν οι ιδιοκτήτες τώρα, ε, βραδία διοικητική διαδικασία ακατάλληλη ή ελλειπής τεκμηρίωση και ε, σύγκρουση συμφερόντων επί της ιδίας περιουσίας και το ζήτημα των προστατευομένων μισθωτών ή ενοικιαστών. Για τη Ρουμανία, εδώ πάλι μιλάμε για διάφορα καθεστώτα ανάλογα με το ακίνητο ε, ή το περιουσιακό στοιχείο. Ε, το 1990 γιατί στα δάση και στις αγροτικές γέες το 90 υπήρχαν κάποια διατάγματα ε, τα οποία έδιναν ε, δικαιώματα σε κάποια μέλη των ε, κολεκτιβών ή συστήματος δηλαδή εκμεταλλεύσεων συλλογικών. Το 1991 ο νόμος για την επιστροφή που προέβλεπε δικαιώματα ε, μετά ε, υπήρχε ένα ανώτατο όριο σε σχέση με τις επιστροφές και καλύφθηκε μόνο η καλύφθηκαν οι γέες που συμπεριλαμβάνονταν σε αυτές τις χειρολογικές εκμεταλλεύσεις. Υπήρχαν και κρατικές εκμεταλλεύσεις που, είχαν, που, ιδιωτικο, που ε, ιδιωτικοποιήθηκαν το 1990. Στο τέλος της δεκαετίας του 90, το 77% των περιουσιακών τίτλων είχαν εκδοθεί καλύπτοντας περίπου το 85% της ε, ε, περιοχής ε, των γεών υπό απέτησης. Τώρα, η περιουσία στη δεκαετία του 90 η μόνη οδός ήταν η δικαστική, ο αστικός κώδικας το 95 το ανώτατο δικαστήριο αποφάσισε ότι αν δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία δεν μπορεί να γίνει επιστροφή. Ε, αυτή ήταν η πρώτη ε, το 1995 είχαμε τον πρώτο νόμο για την επιστροφή εξουσιών με τίτλους, δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει ένας τίτλος ιδιοκτησίας που να έχει δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα που να αναφέρει ότι αφαιρέθηκε, κατασχέθηκε ή απολωτριώθηκε περιουσία και να μπορεί κάποιος να την ζητήσει πίσω. Βέβαια υπήρχαν πάρα πολλές κατασχέσεις χωρίς τίτλο από το κομμουνιστικό καθεστώς. Ε, μπορούσαν επίσης να αγοράσουν οι ενοικιαστές τα διαμερίσματα στα οποία κατοικούσαν. Προβλεπόταν από τον νόμο. Το 1998 ένας νόμος ε, ε, πέρασε για τη δημόσια ιδιοκτησία, ο οποίος πρόβλεπε τη δυνατότητα ανάκτησης περιουσίας από το κράτος, ανεξάρτητα από το πώς έλαβε χώρα η κατάσχεση από το κομμουνιστικό καθεστώς. Όμως δεν υπήρχε πρακτική διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθηθεί αν κάποιος ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο μέχρι το 2001, όταν ε, πέρασε άλλος νόμος για το νομικό καθεστώς των ε, περιουσιών που κατασχέθηκαν από το κράτος που πρόβλεπε και σε είδωσε ε, επιστροφή και αποζημίωση αν δεν γινόταν. Το 2001 διευρύνθηκε το έβρος <clears throat> του νόμου για να καλύψει ακίνητη περιουσία την οποία χρησιμοποιούσε το κράτος για διάφορους σκοπούς, δημαρχία, νοσοκομεία, και τα λοιπά. Και το 2009 ε, ο πρώτος νόμος του 2009 διευκρινίζει ότι η περιουσία που αγοράστηκε από τους ενοικιαστές δεν μπορεί να επιστραφεί σε πρώην ιδιοκτήτες που ε, μπορούν να αποζημιωθούν μόνο. Οι προκλήσεις που βλέπουμε στη Ρουμανία, όπως είπα στην αρχή της παρουσίασης, ε, είχαν σχέση <clears throat> με τις μεγάλες αλλαγές στην συμβολική επιστροφών το πρόβλημα της απόδοσης των, και της καλής λειτουργίας της διοίκησης, γιατί ακόμα κρεμούν πολλά στα δικαστήρια και στη διοίκηση, το ζήτημα των επικαλυπτωμένων δικαιωμάτων και οι διαφορές μεταξύ των ε, ενοικιαστών και πρώην ιδιοκτητών που ζητάνε πίσω τα διαμερίσματα, μακρές διαδικασίες και άνηση δικαστική πρακτική και προβλήματα με το σύστημα των αποζημιώσεων εάν δεν ήταν ε, σε μετρητά, σε χρήμα η αποζημίωση, η χρηματική προβλεπόταν, ε, αλλά για τα υπόλοιπα θα έπρεπε να πάρουν ομολογίες που ακόμα δεν είχαν εισαχθεί στο χρηματιστήριο πράγμα από... και αυτό δημιουργεί πρόβλημα για την πραγματική αξία των ομολόγων αυτών, ομολογιών για τη Σερβία αρχίζω λέγοντας ότι ακόμα δεν έχει ληφθεί απόφαση για τις επιστροφές. Το 2005 θεσπίστηκε νόμος που ζητεί καταχώρηση εθνικοποιημένων περιουσιών και έχουμε εδώ τον αριθμό των αιτήσεων που καταχωρήθηκαν πριν και μετά την προθεσμία. Όμως καμία αίτηση δεν ελέγχθηκε ως προς την ακρίβειά της, στα ακριβή στοιχεία και κανείς δεν γνωρίζει πόσες είναι έγκυρες αν θέλετε. 2002-2003 πρώτο νομοσχέδιο από τη σερβική κυβέρνηση για τις επιστροφές ε, δεν δημοσιεύτηκε ποτέ γιατί το απόσυραν την τελευταία στιγμή. Το 2007 δεύτερο νομοσχέδιο για τις αποεθνικοποιήσεις και αυτό όμως αποσύρθηκε. Το 2009 όμως ε, θε, γκρίθηκε νέος νόμος για το σχεδιασμό και την, τις κατασκευές και μετά υπήρξαν κάποιες εξελίξεις σε σχέση με τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων μεταξύ κράτους και δημοτικών αρχών που εκεί μπορεί να γίνει επιστροφή. Αυτό θα επηρεάσει την επιστροφή όπως και η ιδιωτικοποίηση στη Σερβία θα επηρεάσει τη διαδικασία των επιστροφών. Ευχαριστώ πολύ. Ε, φτάσα στο τέλος της παρουσίασής μου και ευχαρίστω να δεχτούμε ερωτήσεις. Να κάνω μια πρόταση σχετικά με τις εργασίες δεδομένου ότι οι τρεις επόμενες ε, αναφορές αφορούν τις μελέτες ε, που ακούσαμε. Θα δώσω το λόγο στους τρεις ε, αναφέροντες και μετά θα δώσω το λόγο στους βουλευτές που έχουν ζητήσει το λόγο. Αν συμφωνείτε λοιπόν, ούτως θα πράξουμε. Ο κύριος Παραδιάς έχει το λόγο. Thank you very Ευχαριστώ πολύ. Ονομάζομαι στρατό Παραδιάς, ε, δικηγόρος ε, από την Αθήνα και ε, πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτών Ακινήτων. Ακούγοντας τις παρατηρήσεις, τις μελέτες που έγιναν, θα θέλω να πω ότι όταν έπεσε ο τείχος του Βερολίνου προ 20 ετία και όταν πρόσφατα, όταν κατέρευσαν πολλά καθεστώτα στα Παλκάνια οι πολίτες βρήκαν την ελευθερία τους, αλλά πολλοί ε, έμειναν χωρίς τις περιουσίες τους που είχαν κατασχεθεί, απολατρωθεί από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Σήμερα λοιπόν προσπαθούμε να αναλύσουμε ένα πιο περιπλοκό νομικό και κοινωνικό ζήτημα το οποίο άφησαν πίσω τους καθεστώτα τα οποία κατέρευσαν. Συμφωνούμε με τους συντάκτες αυτών των μελετών σχετικά με το ποια, ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες για τη μη επίλυση του προβλήματος μέχρι τούδε. Οι, μελε, μελετητές έκαναν μια πολύ καλή δουλειά. Νομίζω όμως ότι δεν ε, εξέρασαν την περιπλοκότητα του προβλήματος. Βασίστηκαν σε λεπτομέρειες, σε, σε προφορίες μάλλον που τους έδωσαν οι ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις και δεν έλαβαν υπόψη τις απόψεις των θυμάτων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οι μελέτες λοιπόν αυτών, αυτές τείνουν να καταλήξουν ότι ένα τμήμα των προβλήματος έχει σχεδόν επιληθεί κατά ένα ή κατά κάποιο άλλο τρόπο, αλλά είναι, είναι μερικά τα οποία παραμένουν ανεπίλητα. Ξέρουμε ότι πολλές περιουσίες υπάρχουν και μας υπενθυμίζουν αυτήν την πολύ μεγάλη αδικία που υπάρχει. Ε, θα ήθελα να κάνω μερικέ σύντομες παρατηρήσεις για τις χώρες ε, που ακούσαμε. Στην Αλβανία το κράτος ε, δεν αναγνώρισε ότι η διαδικασία για την επιστροφή των ιδιοκτησιών είναι πολύ χρονοβόρος και δαπανηρή. Στην περίπτωση της Βουλγαρίας ε, η μελέτη επικεντρώνεται στο γεγονός ότι οι διοικητικές διαδικασίες που ανέλαβε η κυβέρνηση από το 1991 παρακαλεί τον Μπίλης να διαβάζει λίγο πιο αργά. Η ευκαιρία που έχουν για να τους επιστραφούν οι διοκτησίες τους ε, οφείλεται σε δυσκολίες ε, που δημιουργούν σε διοικητικό και νομικό επίπεδο. Στην περίπτωση της Κροατίας οι μελέτες δεν ασχολούνται με το γεγονός ότι κάποια βασικά έγγραφα ε, παραποιήθηκαν και υπό παράγραφος ε, του άρθρου 3.2 που προβλέπει για την προστασία των δικαιωμάτων από το συνταγματικό δικαίωμα της δημοκρατίας της ε, Κροατίας και αυτό δεν ληφθεί υπόψη. Τώρα, Κάποιες ε, αξίες ε, δεν ε, διχάνουν εγγύηση από, την, από το Σύνταγμα. Στην περίπτωση της Ρουμανίας, Ρουμανίας η καθυστέρηση στην επίλυση του προβλήματος αφορά στην έλλειψη πολιτικής βούλησης και ότι η πιο, φτηνή πιο φθηνός τρόπος για την επίλυση του προβλήματος θα ήταν να επιστραφεί το ακίνητο και να καταβληθούν αποζημιώσεις στον επόμενο ε, ιδιοκτήτη, ο οποίος ήταν και ο αρχικός, ο οποίος είχε αγοράσει την ιδιοκτησία από το κράτος, ο οποίος όμως κράτος δεν ήταν νόμιμος ιδιοκτήτης του ακινήτου. Και τέλος, περίπτωση της Σερβίας, χρησιμοποιήθηκαν πηγές που είτε βρίσκονται υπό το έλεγχο του καθεστώτος ή υπό την ε, πολιτική, τους πολιτικούς ολιγάρχες. Αυτά όλα μας ε, οδηγούν σε λάθος ισχυρισμούς όπως ότι το ε, συμπέρασμα πως μετά από 9 χρόνια εθνικοποίηση στην Σερβία δεν μπορεί να επιβληθεί καμία λύση. Αυτό είναι απολύτως εσφαλμένο και θα πρέπει να δώσουμε στην Επιτροπή σαφή ε, στοιχεία περί αυτού. Καταλήγοντας θα ήθελα να πω ότι μπορέσαμε να ρίξουμε μια ματιά σε αυτές τις μελέτες και επειδή οι ενδιαφερόμενες ε, κυβερνήσεις θα πρέπει να ενημερωθούν από το Κοινοβούλιο, ζητάμε στην Επιτροπή Αναφορών να ζητήσει να γίνει μια περισσότερο σε βάθος μελέτη και να οργανώσει κατά το επόμενο φθινόπωρο εδώ στο Κοινοβούλιο μια συζήτηση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων ε, κρατών με οποιοδήποτε τρόπο εσείς αποφασίζετε έτσι ώστε να εισακουστούν όλες οι γνώμες ε, και όλες οι θέσεις. Εν τω μεταξύ, εκ μέρου τη Διεθνού Ένωση Διοκτών Ακινήτων, σα ζητώ να διατηρήσετε ανοιχτό την, ε, και σε εκκρεμότητα την αναφορά, έτσι ώστε όλοι να κατανοήσουν ότι το Κοινοβούλιο εξετάζει σε βάθο το θέμα και προσπαθεί να, να βρει μια λύση στο πρόβλημα. Ε, Αφήνοντα ανοιχτή λοιπόν την αναφορά μα, ε, θα συνεχίσετε να προσφέρετε ελπίδα που έχει σε άτομα τα οποία έχουν πληγεί και να αναζητηθεί μια νόμιμη και διαρκής λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Κλάουδιος Μότου. Είπε τα βασικά ο κύριος Παραδιά, του δώσα τις ιδέες μου, λέει εκτό μικροφώνου, οπότε δεν θέλω να πάρω το λόγο. Με κάλυψε. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια, στην κυρία Κονσουέλα Φλωρέα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είμαι νομικός και αντιπροσωπεύω τις οκτώ μη κυβερνητικέ οργανώσεις, μεταξύ αυτών και την οργάνωση της οποίας είμαι επικεφαλής. Βρίσκομαι ενώπιόν σα για να σας μιλήσω για τους λόγους που οδήγησαν σοβαρή κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες σύμφωνα με το νόμο 112. Είναι θύματα μιας ε, άδικης ε, διαδικασίας η, νομική ασυνέπεια, η παραβίαση της αρχής της ε, μη της μη οδήγησε στην κατάσταση. Οι επιπτώσεις λοιπόν είναι μια υπόθεση η οποία τελικά έχει καταλήξει ενώπιον του, Ευρωπαϊκού, του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στην περίπτωση λοιπόν της Ρουμανίας δεν λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος με τον οποίο ε, το ζήτημα ρυθμίστηκε σε άλλα κράτη που είχαν ως στόχο να προστατεύσουν τους ε, ενοικιαστές οι οποίοι είχαν αγοράσει από τους ιδιοκτήτες και στις χώρες όπου αποζημιώθηκαν οι πρώην ιδιοκτήτες. Στην έκθεση της Επιτροπής δεν παρουσιάζεται επίσης η περίπτωση των όσων αγόρασαν οι διοκτησίες από την Ρουμανική κυβέρνηση μετά από το 1996, μετά από την εκπνοή της εξάμηνης περίοδου που είχε χορηγηθεί για την υποβολή αιτήσεων. Ε, ο νόμος ε, υπαριθμών 112 εκρίθη συνταγματικός και οι ιδιοκτήτες κατέχουν ένα δικαίωμα το οποίο απέκτησαν μετά το 1994 η ημερομηνία που ε, τέθησε ισχύ τη σύμβαση στη Ρουμανία. Το κράτος ε, έλαβε, εισέπραξε μάλλον πόρους μετά από τις ε, πωλήσει και η κατάσταση που ακολούθησε οδήγησε σε χάος και δημιουργήθηκε ένα σοβαρό πρόβλημα για την επιστροφή των ακινήτων και αυτή που επωφελήθηκε ήταν η, η μαφία που ασχολείται με ακίνητες ιδιοκτησίες. Το δικαστήριο ε, αποφάσισε σχετικά με την υπόθεση Καρακάσου ε, στη Ρουμανία. Αυτή είναι μια υπόθεση η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θεωρούμε ότι το δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο για να εξετάσει τις, ε, την κατάσταση που υπάρχει στον τομέα των διαφορών σε στήματα ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες αγόρασαν τα ακίνητα τηρώντας την ισχύουσα τότε νομοθεσία, δεκαετία του 50. Τα ίδια επιχειρήματα ε, ακούσαμε και από το ε, Συνταγματικό Δικαστήριο της Ρουμανίας στην απόφαση υπαριθμών 73. Θεωρούμε ότι οι επιστροφές έχουν κοινωνικές επιπτώσεις που ξεπερνούν τα όρια μιας εθνικοποίησης. Δεν μπορούμε λοιπόν να αποδώσουμε δικαιοσύνη ε, δημιουργώντας αδικίες. Όσοι λοιπόν κατοικούσαν εδώ και 30 χρόνια σε αυτά τα, σε αυτά τα διαμερίσματα ήταν άτομα τα οποία τελικά εκδιώθηκαν λόγω ε, των αγορών που έγιναν. πολύ πολύ δυστυχώς κατέληξαν στην αυτοκτονία. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θα πρέπει, συγγνώμη, θα πρέπει να λάβουν υπόψη την απόφαση παρθμού 33 της, ε, του Ανώτατου Δικαστηρίου, τον νόμο του 2009, νόμος ο οποίος εκρίθη τρισάκης ε, συνταγματικός και νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια ισορροπία ανάμεσα στους πρώην ιδιοκτήτες και τους νυν ιδιοκτήτες. Χρειάζεται λοιπόν ο νόμος να εφαρμοστεί κατά γράμμα. Μιλάω για το νόμο 2009. Τώρα η ισχύουσα νομοθεσία ε, θα απαιτείται να τροποποιηθεί. Λοιπόν, κάθε αλλαγή όμως τη νομοθεσία δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Η κυβέρνηση της ε, Ρουμανίας θα πρέπει να υποστηριχθεί προκειμένου να μπορέσει να εφαρμόσει την νομοθεσία, νομοθεσία η οποία οδηγεί σε αποζημίωση των ε, προηγούμενων και παλαιών ιδιοκτησιών. Και να πω ότι η Επιτροπή Αναφορών σας ε, καλείται να λάβει υπόψη τις, τις επιπτώσεις ε, κάθε δραστηριότητας ε, σημερινής αλλά και μελλοντική σχετικά με τις επιπτώσεις αναφορικά με την νόμο 112. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Περάσουμε τώρα στους συναδέλφους βουλευτές. Τρεις έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Μποστινάρου. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι των ε, αναφερόντων. Θα ήθελα να αναφερθώ στην έκθεση που αφορά στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που παρουσίασε ο καθηγητής κ. Μπόιτς και θα ήθελα να κάνω τις παρακάτω παρατηρήσεις. Πρώτον, περίμενα η έκθεση αυτή να κάνει αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στην Κροατία σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των προσφύγων και των ε, ενοικιαστών που εγκατέλειψαν ε, τις, ε, τις περιοχές της σύραξης και που σήμερα σύμφωνα με τα στοιχεία του είπα του εκπροσώπου για τους πρόσφυγες μιλάει για, 60, για 70 συγγνώμη, χιλιάδες άτομα άτομα τα οποία προχωρούνται από την Κροατία κατά πλειοψηφία δεν έχουν καμία λύση, δεν τους έχει προταθεί καμία λύση και για να αναφέρω και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προοπτική για την εξέβρεση λύσης θα μπορούσε να είναι ε, να θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και πρέπει να προγραμματοποιηθεί πριν από την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας πω κύριε καθηγητά ότι η δήλωση του Σαράγεβο ε, η συμφωνία του Σαράγεβου, Σαράβι Agreement, είχε ως ε, θέμα την επίλυση του προβλήματος των προσφύγων και των ε, εσωτερικών μετατοπιστέντων προσώπων. Είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό και περίμενα από το Ευρωκοινοβούλιο, το, ως Ευρωκοινοβούλιο μάλλον, το θέμα σας αυτό να θυγεί στην παρουσίασή σας. Τώρα, επίσης, η συμφωνία του Ραμπουγιέ δεν αποτελεί νομικό μέσο. Η συμφωνία του Ρομπουγέ απέτυχε, χρεοκόπησε και ακολουθήθηκε από τον ε, πόλεμο στην Κωσυφοπέριο. Δεν έχει λοιπόν ε, δεν, δεν είναι νομικά δεσμευτικό και η έκθεση Ασιχάρη έγινε δεν μπορεί να γίνει δεκτή διότι ένα κόμμα την απέρριψε. Έχω. Θα ήθελα επίση να σας υπενθυμίσω ότι χώρες όπως η Αλβανία και η Σερβία μέχρι τούδα ε, έχει σχολεία, πολιτικά κέντρα, εκκλησίες και ιδιοκτησίες οι οποίες δεν επεστράφησαν και οι τις δεν υπήρξε καμία αποζημίωση ούτε καν συμβολικού χαρακτήρα. Και εδώ δεν αναφέρομαι για ατομικά δικαιώματα, αλλά μιλάμε για σύμβολα αυτών των οντοτήτων ε, που θα πρέπει να αποτελέσουν ε, θέμα συζητήσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, μελέτη του καθηγητού Στέφαν, να σας πω πως η μελέτη αυτή δεν είναι ε, σωστή καρνάψη των μελών της ε, Επιτροπής μας, διότι η μελέτη αυτή δεν ε, ασχολείται με την διαχείριση αυτού του τραγικού φακέλου για την ιστορία των πρώην κομμουνιστικών χωρών και αναμειγνύει πράγματα άσχετα μεταξύ τους. Δεν θα πρέπει λοιπόν να μπλέκουμε μελέτες που αφορούν στη Ρουμανία και την Βουλγαρία με μελέτες που αφορούν ε, χώρες ε, που προσβλέπουν στην ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχουν κάποιες κατευθύνσεις γραμμές που μπορούν να μας βοηθήσουν με τέτοιου είδους μελέτες. Δεν υπάρχει συνεκτικότητα και αφετέρου δεν γίνεται αναφορά σε περιπτώσεις ε, που ε, στέφθησαν από επιτυχία και που είχαν θετικότατα αποτελέσματα όπως βέβαια της Γερμανίας, της Τσεχίας, της Σλοβακίας, της Ουγγαρίας. Χάρη λοιπόν στις χώρες αυτές λάγω της ε, σαφήνειας ε, του νομοθέτη οι επιπτώσεις ε, ήταν ελάχιστες. Η μελέτη λοιπόν δεν θίγει διόλου αυτές τις πτυχές και δεν αναφέρει το τι θα πρέπει να κάνουν τα κράτη των Βαλκανίων για να μην υποπέσουν στα ίδια σφάλματα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι ο ρόλος παρομοιών μελετών και κάτι ακόμα. Περίμενα η μελέτη σας να κάνει τουλάχιστον μία αναφορά στα θέματα της ε, σοβαρής διαφθοράς που έχουν εμπλακεί σε ό,τι αφορά την επιστροφή των ε, περιουσιών και των ιδιοκτησιών. Η ε, μαφία που δράστονται με τον των ακινήτων και η διαφθορά του νομικού συστήματος οδήγησε σε αποφάσεις πραγματικά απαράδεκτες οι οποίες ε, είτε επικυρώθηκαν είτε βρίσκονται ακόμα ενώπιον της δικαιοσύνης. Και σε ό,τι φορά την τελευταία αναφορά των ε, Ρουμάνων αναφερόντων την υποστηρίζω ε, και εδώ δεν είμαστε δικαστήριο, είμαστε πολιτικοί άνδρες και γυναίκες και σας ερωτώ κύριοι συναδέλφοι, μπορούμε να δεχτούμε σε ένα μέλος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύο εκατομμύρια άτομα να, να χάσουν το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και να κινδυνεύουν να βρεθούν στο δρόμο όπως σας είπα, υπήρξαν αυτοκτονίες. Πρόκειται για μια κατάφορη αδικία του κομμουνιστικού καθεστώτος, αλλά που σήμερα καθιστάται από μια ακόμα αδικία του κοινωνικού και του οικονομικού συστήματος. Και κάτι ακόμα. Δεν πιστεύω ότι κράτος Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να δεχθεί δύο εκατομμύρια των πολιτών του να απειλούνται να βρεθούν στον δρόμο διότι με διαφορά σχέση με την Γερμανία, την Πολωνία, την ε, Τσεχία και άλλα κράτη δεν υπήρξε δυνατότητα για τους ενοικιαστές που εν τω μεταξύ έγιναν ιδιοκτήτες ε, να αποκτήσουν ένα, ένα συμβόλαιο Πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν ηλικία 70-75 χρόνια και δεν μπορούν να ανακτήσουν τις περιουσίες τους ε, και αυτοί θα είναι τα πραγματικά θύματα της όλης διαδικασίας ε, και θα ολοκληρώσω εδώ παρακαλώντας σας ε, να τα λάβετε όλα αυτά υπόψη η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δεχτεί δύο εκατομμύρια άνθρωποι να αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα και να μην δείχνουμε καμία συμπόνια από εμείς ως κράτη-μέλη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 Συγγνώμη, με συγχωρείτε, να ξαναρχίσω. Έλεγα λοιπόν ότι επιθυμώ να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, γιατί ήθελα να ε, είμαι ακριβή στη διατύπωση. Να συγχαρώ για τις μελέτες εμβαθύνατε στο θέμα, το οποίο εξακολουθεί μέχρι σήμερα να είναι πολύ ευαίσθητο. Τρεις σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτον, με τα, τα μέτρα. Γιατί δεν βλέπετε τις χώρες που δεν επικεντρώνεστε στις χώρες που τώρα είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παλιά ήταν κομμουνιστικές όπου η ιερότητα της ατομικής ιδιοκτησίας είχε ε, παράφορα καταβιαστεί με ένα σωρό απαλωτριώσεις, σχέση κλπ. Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία. Σε αυτές τις χώρες λοιπόν βλέπουμε ακόμα τις συνέπειες του προπατορικού κομμουνιστικού αμαρτήματος Ακόμα έχουμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα και παρόμοια είναι τα πράγματα σε αυτές τις χώρες και στη συμπανάληση ε, από εσάς χώρες. Ένα παράδειγμα για να δείτε πόσο δύσκολο πρόβλημα ηθικό είναι αυτό. Ο Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας μέχρι σήμερα ζει σε μία βίλα η οποία ε, αφαιρέθηκε από μια εβραϊκή οικογένεια από τους Ναζί και μετά για δεύτερη φορά παλωτριώθηκε από τους κομμουνιστές και ο κύριος ο Πρωθυπουργό δεν ενοχλείται που μένει σε αυτή τη βίλα Αυτές είναι οι αμαρτίες οι παλιές που εξακολουθούν να μας ε, ταλανίζουν και σήμερα. Γιατί λοιπόν να μην δούμε τι γίνεται και σε αυτές τις χώρες, γιατί δεν τις συμπεριλάβατε στη μελέτη σας. Δεύτερο, είχα την εντύπωση ότι κανένας από τους συντάκτες, καθηγητές, δεν κάνει σαφή διάκριση μεταξύ αποζημίωσης και επιστροφής, παρόλο που πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Η αποζημίωση στην Ουγγαρία έγινε με τη βοήθεια αυτών των ομολόγων, κάτι κουπόνια, vouchers. Αυτό ήταν άδικο. Ήταν μια φθηνή ε, μέθοδος. Αυτά μπορούσαν να πολιθούν, αλλά και αργότερα ποτέ δεν θεωρήθηκαν πραγματική αποζημίωση. Η επανιδιωτικοποίηση, η οποία αναφέρθηκε από τους ομιλητές, ως εάν ήταν μια μορφή επιστροφής, από ό,τι γνωρίζω δεν αποτελεί επιστροφή. Δεν έγινε επιστροφή. Στην Ουγγαρία σίγουρα όχι. Δεν έγινε επιστροφή. Και από ό,τι ξέρω και σε άλλες χώρες δεν έγινε. Δηλαδή ε, ούτε καλλιεργούμενες γιές ούτε ακίνητα, ούτε ε, κίνητα επεστράφησαν. Και αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο γιατί ακόμα έχουμε να αντιμετωπίζουμε αυτή την ανηθικότητα αν θέλετε. Υπήρξαν κάποιες προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί το ηθικό αυτό πρόβλημα με αυτές τις, ε, μετά από αυτές τις ε, φαινομενικές ε, αποζημιώσεις να περάσουν σε γνήσια αποζημίωση, επιστροφή δηλαδή. Οι Ναζί και οι κομμουνιστές απαλωτρίωσαν πάρα πολλές περιουσίες και υπήρξε εδώ μεταξύ αλυσίδα διαφορετικών ιδιοκτητών που μεσολάβησαν. Αν επιστραφεί τώρα η ιδιοκτησία, η περιουσία, θα αδικηθεί και θα απαλατριωθεί, αν θέλετε, ο εντωμεταξύ νόμιμος ιδιοκτήτης Δηλαδή, εννοώ ότι δεν μπορούμε μια αδικία να την ε, ε, βελτιώσουμε και να την αντιμετωπίσουμε με μια δεύτερη αδικία. Ενδεχομένως ε, θα υπήρχε μια πρακτική, νομική αλλά και ηθική μέθοδος για την αντιμετώπιση του δύσκολου προβλήματος της επιστροφής. Ευχαριστώ συνάδελφος Μακμίλαν, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ ενδιαφέρομαι από χρόνια για αυτό το θέμα. Ήμουν από τους πρώτους εισηγητές της Επιτροπής Αναφορών για διασυνοριακά θέματα ιδιοκτησίας το 1998. Και ευχαριστώ την Επιτροπή και τα προηγούμενα μέλη που ανέθεσαν αυτές τις μελέτες και το προσωπικό που τις ετοίμασε τις μελέτες και στα διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Το θέμα που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το εξή. Είναι πολύ ευρύ το θέμα. Επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπου σε όλη την Ευρώπη. Αυτό υπόθηκε όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στι υποψήφιε χώρε και ενδεχομένω και άλλε. Και γι' αυτό νομίζω ότι δεν θα πρέπει να αφήνουμε εδώ αυτά τα θέματα και μόνο. Να τα σταματήσουμε. Το θέμα των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας για πρώτη φορά συζητήθηκε στα πλαίσια του άρθρου 17 στο ΔΕΚ όσον αφορά τα τρέχοντα δικαιώματα και αυτό δεν επηρεάζει απαραίτητα τα προϋπάρχοντα δικαιώματα και αυτό σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να έχει μια συνεχτική θέση όσον αφορά τα θέματα ιδιοκτησίας εν γέννη και υπάρχουν πάρα πολλά και περίπλοκα ζητήματα που τίθενται εδώ και αλλαχού. Λοιπόν, το εξή έχω να πω κύριε Πρόεδρε, ας μην σταματήσουμε εδώ. Το άλλο που έχω να πω είναι πιο συγκεκριμένο. Ξέρω αρκετά για τα όσα συμβαίνουν στη Σερβία. Ε, πήγα εκεί πιο πολλές φορές από τις άλλες βαλκανικές χώρες. Δεν πιστεύω πραγματικά ότι η έκθεση με κάθε σεβασμό καλύπτει επαρκώς το θέμα της διαφθοράς, της κολυσιεργίας. Το θέμα των δυσκολιών για τους νόμιμους ιδιοκτήτες όταν προσπαθούν να επιδιώξουν επιστροφή. Τίποτα δεν έχει συμβεί, τίποτα. Τίποτα δεν έχει συμβεί στη Σερβία. Και επειδή θέλει να γίνει και μέσω Ευρωπαϊκή Ενώσεω, θα πρέπει να προσέξουμε όλου ιδιαίτερα σε αυτό το θέμα, λαμβάνοντα υπόψη ότι η Συμφωνία Σερβία με την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται συγκεκριμένα στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Μέσω ημών, κυρία Πρόεδρε, διερωτώ με μήπω θα ήταν δυνατόν η Επιτροπή Αναφορών να διορίσει έναν εισηγητή μέσω των συντονιστών. Σκεφτείτε το. Ή εν γέννη, βλέποντας τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που επηρεάζει ιδιαίτερα αυτή την Επιτροπή και τα δικαιώματα των παιδιών. Αυτά είναι συμπληρωματικά θέματα και ετοιμάζεται άλλη μελέτη γι' αυτό. Θα έλεγα να γίνει μια κοινή ακρόαση αργότερα φέτο, να καλύψουμε τα δύο θέματα, τα δικαιώματα των παιδιών και τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Είναι οι δύο νέε πτυχέ τη συνθήκη της που αποτελούν θεά ζώνη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θεμητό ενδιαφέρον για αυτό το θέμα. Από ό,τι ξέρω, αν σταματήσουμε εδώ, λησμονούνται τα θέματα. Και ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο αυτό το ζήτημα που συζητούμε. Πέρσι έγινε μια δήλωση για την επιστροφή ε, ε, περιουσιών προπολεμικών. Επικυρώθηκε από 40 χώρες. Επιστροφή κυρίως σε εβραϊκές οικογένειες ε, παλαιών περιουσιών. Υπάρχουν πολλοί βουλευτές που ενδιαφερόταν, δεν είναι εδώ σήμερα. Θα ήθελαν να υπάρχει ένας πιο διεκπαιρωτικός μηχανισμός, όπως μια κρόση από τη μια συνάντηση Επιτροπή. Έκκληση απευθύνω να παραμείνει ανοιχτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Πασέσκου. Ε, κυρία Πασέσκου. Ευχαριστώ. Το ίδιο σχόλιο όπως και συνάδελφος Έχω εγώ σχόλια γιατί η Ρουμανία και η Βουλγαρία συμπεριλαμβάνονται στην ίδια μελέτη με τις Βαλκανικές χώρες. Διότι η Ρουμανία και η Βουλγαρία είναι ήδη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεω Σε πιο προθυμένα στάδια αντιμετωπίσεω του θέματο της επιστροφής των περιουσιών. Θέλω να προβώ στα κάτω σχόλια. Όσον αφορά τις αναφορές του κ. Βιτζίστερε και θα αναφερθώ σχετική νομοθεσία. Οι πρώην ιδιοκτήτες περιουσιών που κατασχέθηκαν από το κράτος κατά το κομμουνιστικό καθεστώς και το καθεστώς εκείνων που κατοικούν στα ε, κτίρια αυτά καλύπτονται παράλληλα. Οι ρουμανικές αρχές ήθελαν να εξασφαλίσουν ισότιμη αντιμετώπιση και μη διάκριση μεταξύ δύο κατηγοριών. Ε, απ' τη μια, εκείνους που ήταν αντικείμενο καταχρηστική μεταχείρισης από τη μια πλευρά και από την άλλη ε, έχουμε εκείνους τους οποίους το κράτος έδωσε την διοκτησία μετά. Ο κ. Καταλήν Πεντογιού, Ρουμάνο Υπουργό Δικαιοσύνη, απάντησε στην αναφορά σε επιστολή που παρουσίασε Ακροθυγός ε, την ρουμανική νομοθεσία. Και τώρα σα παρουσιάσω την νομοθεσία. Νόμο υπαριθμών 112 είναι η πρώτη πράξη που έδωσε στους πρώην ιδιοκτήτες τη δυνατότητα να ζητήσουν επιστροφή των σπιτιών τους που κατασχέθηκαν καταχρηστικά από το κράτος. Ο ίδιος νόμος παρήχε τη δυνατότητα στους μισθωτές βάσει αυτών των συμφωνιών να αγοράσουν τα σπίτια. Λοιπόν, έχουμε τον νόμο 10.2001. Οι πρώην ιδιοκτήτε ιδιοκτησιών που κατασχέθηκαν από το κράτο κατά το κομμουνιστικό καθεστώ μπόρεσαν να ζητήσουν επιστροφή ή αποζημίωση εις είδος ως ενδείκνεται. Τα κενά κτίρια επιστρέφονται στους πρώην ιδιοκτήτες εις είδος. Στην περίπτωση που δεν καταργήθηκαν κατά συμβόλαια πωλήσεως κτηρίων ή των κτηρίων των αδείων οι διοκτήτε ή κληρονόμοι δέχθηκαν απλώ αποζημήωση. οι κληρονόμοι δέχτηκαν απλω αποζημίωση. Η επιστροφή ειδο είδος αποκλείεται τη αυτή περιπτώση. Είναι απαραίτητο το δικαστήριο να καταργήσει τη σύμβαση πωλήσεω μέσω τελεσίδικης απόφαση, ώστε ο πρώην ιδιοκτήτη να δεχτεί σε επιστροφή την περιουσία που ε, πολίθηκε στον μισθωτή. Ο νόμος 10 του 2001 τροποποιήθηκε και ολοκληρώθηκε από το νόμο 1 του 2009 ο νόμος 10 του 2001 τονίζει ότι οι πρώην ιδιοκτήτες σύμφωνα με τον νόμο 112 των οποίων οι συμβάσεις πωλήσεων ακυρώθηκαν από την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου πρόκειται να λάβουν είτε αποζημίωση που αντιπροσωπεύουν την πραγματική αξία αγοράς του κινήτου ή την τιμή αγορά σύμφωνα με το δίκτυ τιμών ο κ. Πρεντόγιο, Υπουργό Δικαιοσύνη, εξέδωσε την εντολή παριθμών 40 του 1999 που αφορούσε σύστημα εγγύσεων για τους μισθωτές και για τα δικαιώματά τους και για να εξασφαλιστεί στέγαση από εκείνους που εκδιώχθηκαν από τη χρήση προστάσεων στους πρώην ιδιοκτήτες είχαμε το διάταγμα 74 της κυβερνήσεως του 2007. Όλες αυτές οι πράξεις είχαν σαν στόχο να αποζημιώσουν τις καταχρήσεις του κομμουνιστικού καθεστώτος και να παράσχουν την καλύτερη δυνατή κοινωνική προστασία. Για να αποζημιωθούν οι πρώην ιδιοκτήτε, πρέπει να γίνει και αντιστάθμιση και με τα συμφέροντα εκείνων που μένουν. Ο, ο νόμος 10 του 2001 επικυρώθηκε αφού το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάσισε ότι συνάδει με το Σύνταγμα. Ήθελα να σας πω ότι έχουμε νομοθεσία σχετικά με το ζήτημα. δεν ήθελα όμως να καταλήξω σε κάποια κρίση και σε κάποιο πόρισμα, σε κάποια απόφαση. Πώς να παρουσιάσω την εικόνα ήθελα. Κύριε Ράπτη. άκουσα με πολύ προσοχή όλους τους ομιλητές. Ε, η κατάσταση δεν είναι καθόλου απλή. Είναι, θα έλεγα, περιπεπλεγμένη, περίπλοκη και κρίσιμη. Ε, μέσα σε όλα αυτά και για να μπορώ να έχω ένα περισσότερο ξεκάθαρο ε, τοπίο, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον πρόεδρο στον εκπρόσωπο της Διεθνούς Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων, στον συμπατριώτη μου κύριο Παραδιά. Ε, θα ήθελα να επαναλάβει, ε, να τον ακούσω να επαναλαμβάνει τις χώρες που αφορά, έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό και σαφές, εντελώς σαφές, ότι αυτή η ιστορία αφορά α, περιπτώσεις περιουσιών μέσα στο ίδιο κράτος και όχι από ένα κράτος σε άλλο. Ε, θα ήθελα αυτή τη διευκρίνηση από τον κύριο Παραδιά. Ε, τελειώνω πάρα πολύ σύντομα ε, λέγοντας το εξής. Με τα όσα έχω ακούσει με πολύ προσοχή από όλους τους ομιλητές, ε, θα ήθελα δύο πράγματα. Πρώτον, ε, οι μελέτες μου φαίνονται λιγάκι επιτρέψτε μου τον όρο χαοτικές. Δηλαδή θα τις ήθελα από μία μελέτη, περιμένω να είναι περισσότερο ε, μεθοδολογικά δομημένη. Και βέβαια θα βοηθούσε πολύ περισσότερο εάν μπορούσαμε να είχε ο κάθε βουλευτής ένα αντίτυπο αυτής της μελέτης, ώστε πραγματικά να έχουμε το χρόνο να μελετήσουμε διεξοδικά ένα τόσο σοβαρό ζήτημα από μια σύντομη παρουσίαση που όντως οι παρουσιαστές έκαναν κάθε προσπάθεια να την κάνουν εύκολα αντιληπτή ε, δεν είναι δυνατόν να, να εξαντληθεί το θέμα. Άρα το ένα ζήτημα είναι ότι θα ήθελα εγώ τουλάχιστον να έχω στο χέρι μου ε, μία περίληψη, μία σύνοψη των μελετών ώστε να μην αδικήσω ενδεχομένως και τους ανθρώπους που έκαναν την έρευνα. Θέλω να είμαι δίκαιη, αλλά δεν μου δίνουν αυτή τη στιγμή ε, το εργαλείο για να είμαι ε, αντικειμενική. Άρα θέλω περισσότερη ενημέρωση. Ένα ζήτημα αυτό. Και δεδομένων των καταστάσεων που επικρατούν, ε, θα ήθελα, αισθάνομαι ότι θα ήθελα να μείνει το ζήτημα ανοιχτό. Δεν πρέπει να κλείσει ακόμη, κατά τη γνώμη μου, γιατί ε, έχει να γίνει ακόμη πολλή συζήτηση και να διευκρινιστούν πολλά ζητήματα. Grazie, Presidente. Ο κύριε Πρόεδρε, ε, σαν μελέτες όπως τις άκουσα και σαν νομικός που είμαι, θεωρώ ότι αποτελούν ε, μια περιληπτική ενημέρωση του σώματος σχετικά με το πρόβλημα των ιδιοκτησιών στα τέως ανατολικά κράτη, στα τέως κομμουνιστικά κράτη που υπήρξαν στα Βαλκάνια. Και λέω στα τέως κομμουνιστικά κράτη που υπήρξαν στα Βαλκάνια, διότι δεν ήταν όλα τα κράτη των Βαλκανίων κομμουνιστικά. Υπήρχε και η Ελλάδα, μια ελεύθερη χώρα, η οποία ε, δεν έχει καμία σχέση με αυτά ε, τα οποία συμβαίνουν στις τέσσερις ανατολικές χώρες συμμερίζεται βεβαίως το πρόβλημα το οποίο υπάρχει για τους ανθρώπους που ζουν σε αυτές και, είναι, και κατάγονται από αυτές. Ε, βεβαίως, στα πλαίσια της ενημερώσης μιας επιτροπής που δεν έχει δικαστικό χαρακτήρα, γιατί δεν είμαστε δικαστήριο εδώ, είμαστε μια επιτροπή η οποία βλέπει το κοινωνικό κυρίως στοιχείο του προβλήματος, νομίζω ότι χρειάζεται μια συμπλήρωση των μελετών αυτών ε, και συμφωνώ με την κυρία Ράπτη ότι καλό θα ήταν να τις έχουμε προηγουμένως και να τις μελετήσουμε διότι καθώς αντιλαμβάνεστε ε, συμπλέκονται πολλές διατάξεις δικαίου. Συμπλέκονται διατάξεις συνταγματικού δικαίου, συμπλέκονται διατάξεις εμπραγμάτου δικαίου, συμπλέκονται θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, συμπλέκεται και το θέμα της πορείας των χωρών αυτών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι συμφωνώ με τον κύριο Μποστινάρου ότι δεν έχουμε την ίδια πορεία στις χώρες που ήδη είναι ενταγμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την αποκατάσταση τη δημοκρατία, διότι θεωρώ και είναι αποκατάσταση τη δημοκρατία η επιστροφή των περιουσιών, αφού όλα τα δημοκρατικά συντάγματα, από τη Μάγνα Χάρτα του 1215 έω το Ζάξεν Σπίγκελ του 1400 του Γερμανικού, περιέχουν διατάξει περί Συνεπώ, η αποκατάσταση στις λειτουργίες της δημοκρατίας στις χώρες αυτές που είναι ήδη ενταγμένες ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι είναι επαρκέστερη και εν πάση περιπτώσει σε καλύτερη μοίρα από ό,τι στις άλλες χώρες ε, οι οποίες αναφέρθησαν στις συγκριτικές μελέτες και οι οποίες ε, ε, μας δόθηκαν με γλαφυρό τρόπο οφείλω να πω από τους συναδέλφους μου νομικούς. Όμως πρέπει να μείνει, συμφωνώ ότι πρέπει να μείνει ανοιχτή το όλον θέμα με την διευκρίνηση ε, ότι δεν αφορά την Ελλάδα, το λέω αυτό, διότι μην ξεχνάμε ότι τα Βαλκάνια είναι μια χώρα στην οποία υπήρξαν πολλές δικαιοδοσίες και πολλοί πολιτισμοί. Υπήρξε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία με δικό της δίκαιο το οποίο αναφέρθηκε. Και αναφέρθηκε εμέσως διότι υπήρξε το, το τουρκικό υποκατάστατο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το οποίο είχε διατάξει σε πραγμάτου δικαίου οι οποίες εφαρμόζονται σε πολλές από τις χώρες αυτές και υπήρχε ιδιαίτερα στις ε, γειτονικές χώρες προς την Αυστρία και Γερμανία. Ε, το είδαμε στην, ε, ε, στην χώρα, την, την Βοσνία και την Ερζεγοβίνη που έχουν περισσότερο διατάξει ευρωπαϊκού δικαίου παρά διατάξεις Οθωμανικού δικαίου που έχουν τις ρίζες τους και αυτές στο παλιό Βυζαντινό δίκαιο, το οποίο και αυτό στο παλιό Ρωμαϊκό δίκαιο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν με το κομφούζιο το οποίο υπάρχει στην περιοχή εάν δεν διευκρινίσουμε ότι αφορά αποκλειστικά η όλη υπόθεση τις χώρες τις τέως ανατολικές που υπέστησαν αυτό που υπέστησαν με τον κομμουνισμό, καλός ή κακός αυτός ήταν, με αυτόν έζησαν και τις συνέπειες αυτού πληρώνουν ή δεν πληρώνουν διότι υπάρχουν πολλές απόψεις, ο καθένας έχει τις πολιτικές που τις οποίες σέβομαι σε αυτό θα ήθελα να έχουμε μια ενημέρωση για μελλοντική συνάντησή μας ε, έγγραφοι σχετικά με τις απόψεις των μελετητών για να είμαστε σε θέση να πούμε και περισσότερα πράγματα και ουσιαστικότερα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να διευκρινίσω πως τα κείμενα διανεμήθηκαν εδώ και δύο εβδομάδες, αλλά όσοι τα εζήτησαν εκ νέου σήμερα θα φροντίσω να σας διαβιβαστούν. Το λόγο έχει εκπρόσωπος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπατε ήδη σχετικά με την αποδυναμωμένη αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρέπει να πω ότι οι κανόνες δεν έχουν αλλάξει. Δηλαδή δεν υπάρχει διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη απάντησή μας στις αναφορές. Ό,τι είπαμε ισχύει. Η βάση μας για ανάληψη δράσης είναι τα κριτήρια προσχώρησης, ένταξης. και όταν πρόκειται για προστασία δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, ε, αυτό ε, είναι ενσωματωμένο στα κριτήρια ένταξης. Οι επιστροφές πρέπει να στηρίζονται στην εθνική νομοθεσία, αλλά πρέπει να γίνονται και με τρόπο δίκαιο και διαφανή και με πλήρη σεβασμό του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επίσης σημαντικά είναι όλα αυτά και για τα οικονομικά κριτήρια ένταξης. Όταν ας πούμε υπάρχει διοκτησία ακινήτων που δημιουργεί εμπόδια για τη λειτουργία της αγοράς και ε, είναι εμπόδιο στα, κριτήρια, στα οικονομικά κριτήρια ένταξης. Επίσης οι διακρίσεις στην ιδιοκτησία κινήτων δημιουργεί πρόβλημα στις ε, ε, εθνικές και ξένες επενδύσεις, στην παραγωγικότητα και γενικότητα της γεωργία και γενικά. Ε, θεμελιώδες επίσης για τη λειτουργία της αγοράς. Είναι να διασφαλίζονται δικαιώματα ε, ακινήτων τα οποία βεβαίως θα μπορούν μετά να αποτελούν τη βάση και για ενυπόθηκα δάνεια, ε, δάνεια για επενδύσεις κλπ. Να πω δύο λόγια και για την πρόσφατη εξέλιξη στην επιστροφή περιουσιών στο Κωσυφοπαίδιο και στα Δυτικά Βαλκάνια γενικότερα. Στη Βοσνία Ερζεγοβίνη δεν υπάρχει σαφές νομικό πλαίσιο ακόμα. Σε κρατικό επίπεδο οι καθυστερήσεις προέρχονται από την αντίσταση κάποιων πολιτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης που αμφισβητούν την κοινοβουλευτική συνέλευση και την άρμο εξουσία που έχει να νομοθετεί για επιστροφές μεταξύ άλλων περιουσιών. Υπάρχουν προβλήματα με την δημοκρατία της Σερβίας που διαφοροποιείται στις επιστροφές. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για βιώσιμη και εναρμονισμένη λύση. Ακούσαμε και τα προβλήματα στην Κροατία. Οι εκρεμείς υποθέσεις επιστροφών και αποζημιώσεων. στηρίζεται στη νομοθεσία των αρχών του 90, αλλά εξακολουθούν να εκρεμούν στην Σερβία δεν υπάρχει νομική βάση, οπότε δεν μπορεί να αρχίσει όπως πρέπει και η διαδικασία των επιστροφών. Η ιδιωτικοποίηση ε, συνέχισε με κάποιους κινδύνους σε σχέση με την αντιμετώπιση των επιστροφών. Μετά την οικονομική κρίση και τους στενούς προϋπολογισμούς η διαδικασία αντιμετωπίζει ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις. Για το κοσυφοπαίδιο, εκεί η κατάσταση ακριβώς περιεγράφει στις μελέτες. η ε, ε, περιουσιών υπεύθυνο για την αντιμετώπιση των επιστροφών, αλλά τελική απόφαση θα ληφθεί από τα δικαστήρια, από τις δικαστικές αρχές. Ο φορέας αυτός έχει ενισχυθεί οικονομικά και η Σερβία και το Κωσυφοπαίδιο πρέπει να συνεργαστούν οπωσδήποτε για να λύσουν περιουσιακά θέματα. Αλλιώς δεν θα υπάρξει σημαντική πρόοδος, βράχη πρόθεσμα. Σωστά συμπεραίνουν οι μελέτες ότι η επιστροφή περιουσιών είναι σημαντική για τη διαδικασία επιστροφής γενικότερα η διαδικασία του Σαράγεβο δυστυχώς δεν έδωσε καρπούς τους αναμενόμενους τουλάχιστον ε, μετά την, όπως διαπιστώθηκε στην Υπουργική Σύνοδο 25 Μαρτίου. Οπότε είναι μπλοκαρισμένη η κατάσταση μεταξύ χωρών. Εμείς στηρίζουμε ε, τις προσπάθειες διευκρίνησης περιουσιακών θεμάτων στη, στα προγράμματα, για παράδειγμα, κατα, ε, καταχώρησης περιουσιών στα κτηματολόγια. Ευχαριστώ. Να, δώσω τώρα το λόγο για δύο λεπτά από, σε κάθε, από τους αναφέροντες. Δύο λεπτά ο καθένας. Κύριε Μικρόφωνο παρακαλούμε. Σύντομη δήλωση για να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Η αναφορά η συγκεκριμένη αναφέρεται στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα περιουσιών που κατασχέθηκαν από κράτη που ήταν στο παρελθόν υπολοκληρωτικά καθεστώτα. Ο κομμουνισμός ήταν τέτοιο καθεστώς, ο φασισμός ήταν τέτοιο καθεστώς. Αναφερόμαστε ακριβώς σε αυτό. Και αναφερόμαστε σε αξιώσεις πολιτών ευρωπαϊκών χωρών κατά των ιδίων τους χωρών. Ρουμάνοι που ζητάνε επιστροφή περιουσιών από τη Ρουμανία. Βούλγαροι που ζητούν επιστροφή ιδιοκτησών από τη Βουλγαρία. Δεν μιλάμε για Ρουμάνους που ζητούν περιουσίε από τη Βουλγαρία. Η οδήποτε αξίωση από χώρε που ποτέ δεν είχαν ολοκληρωτικό καθεστώ. Όπω η Ελλάδα ποτέ δεν είχε τέτοιο καθεστώ. Είναι ξεκάθαρο τι αφορούν αυτές οι αξιώσεις για ιδιοκτησίες ακινήτων και τι υποστηρίζουμε. Δεν υπάρχει ουδέμια αμφιβολία Ακριβώς αυτό αναφερόμαστε. Ευχαριστώ. Grazie. Σας ευχαριστώ. Ακολουθούμε τη σειρά που ακολουθήσαμε πριν όσον αφορά τους ειδικού. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή που είναι ευρύτατη όπως άλλωστε και η θεματική μας. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, γι' αυτό ζητώ την κατανόησή σας. Εμείς είμαστε νομικοί και η προσέγγιση μας καμιά φορά είναι διαφορετική από τη δική σας. Προσπαθήσαμε και υπήρχε μια ένσταση γιατί η Βουλγαρία και η Ρουμανία συμπεριλήφθησαν εδώ. Αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα γι' αυτό. Εμείς ε, ε, δουλέψαμε πάνω στις χώρες ε, ε, που μας ανέθεσαν να εξετάσουμε και να μελετήσουμε. Προσπαθήσαμε να κάνουμε διαφοροποίηση όμως, να δούμε τη διαφορετική διάσταση, δηλαδή τις υποχρεώσεις του κράτους μέλους, ε, τις υποχρεώσεις του κράτους μέλους που είναι σε ένα άλλο στάδιο, σε στάδιο το οποίο ε, επιδιώκει την εναρμόνιση και το Κωσυφοπέδιο και η Σερβία που απέχουν ακόμα από όλα αυτά. Η διαφοροποίηση ήταν πολύ σημαντική και έγινε από εμά. Άρα λοιπόν ε, μιλάμε για διαφορετική βαθμίδα ανάπτυξης και ε, δεν τα βάλαμε όλα σε ένα τσουβάλι. Αυτό θέλαμε οπωσδήποτε να το αποφύγουμε. Τώρα, για την επανειδιωτικοποίηση, καρποτλάζ στην θεωρία ε, ξισούται με την αποζημίωση και το reprivatizatio με την επιστροφή. Δηλαδή, καμιά φορά είναι θέματα ορισμών, ετοιμολογίας, αλλά πάντως έχετε δίκιο ότι η διαφοροποίηση θα πρέπει να γίνεται με πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Αλήθεια είναι αυτό. Επίσης, ε, πόσο πίσω θα πάμε. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε ως επιτοπλίστων θα πρέπει να δούμε από το 45 τα πράγματα. Ε, μπορούμε να πάμε και πιο πίσω όμως, ανάλογα. Μπορούμε να εξετάσουμε και άλλες περιόδους. Αλλά αυτά είναι θέματα που κρίνονται πολιτικά και αποφασίζονται, δεν είναι νομικά. Ο νομικός καλείται να απαντήσει στα ερωτήματα που του θέτει ο πολιτικός. Το λόγο έχει ο αναφέρον Μόρτ, τον οποίο δεν είχα δει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να πω καταρχήν ότι τα δύο εκατομμύρια θύματα, ότι ο αριθμός αυτός είναι πολύ εντυπωσιακός, αλλά δεν είναι αληθής, δεν είναι ακριβής. 200.000 αιτήσει κατατέθηκαν στη Ρουμανία και από αυτές τις 200.000 οι περισσότερες αφορούν ε, αγροτικές γέες, ε, ε, αγροτικά αγαθά. Μπορεί να είναι 500.000 για γέες το πολύ και 2 εκατομμύρια θύματα. Λέει πώς καταλήξατε σε αυτό το ποσό, σε αυτό τον αριθμό. Δεύτερον, να υπενθυμίσω ότι οι κατασχέσεις από το 1950 ε, έγιναν παραβιάζοντας την τότε ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή και τότε διεπράχθη αδίκημα. Και τότε είχε διαπιστωθεί η παράβαση. Εκείνη την εποχή το κράτος είχε αποκτήσει τίτλους ιδιοκτησίας που δεν είναι δικαιούτο να έχει. Και αυτό δεν είναι γνώμη δική μου μόνο, είναι μια διαπίστωση την οποία έκανε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που σε μία απόφαση είπε ότι πώλησε, επόλυσε τίτλους στο κράτος που δεν του ανήκαν. Επίσης, ο, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνέστησε στο Ρουμανικό κράτος το ταχύτερο δυνατόν να θεσπίσει μέτρα ώστε οι ιδιοκτήτες που τους απαλωτρίασαν την ε, περιουσία τους ή ε, να επιστραφεί ή να αποζημιωθούν το ταχύτερο δυνατό. Το ταχύτερο δυνατό αποζημίωση. Αυτή η διατύπωση είναι του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο δικαστήριο ε, άρχισε μια διαδικασία πιλωτική Μία διαδικασία, μία προσφυγή θα γίνει τον Ιούλιο κατά της Ρουμανίας, ε, πρότυπο δηλαδή, και θα πρέπει να ε, αποζημιώσει ή να επιστρέψει η Ρουμανία. Επίσης, η Υπουργική Σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 4 Μαρτίου φέτος, στην 1708, ε, ζήτησε από τη Ρουμανία να λάβει μέτρα ούτως ώστε οι συστάσεις αυτές να εφαρμοστούν στην πράξη. Να υπενθυμίσω και κάτι ακόμα. Συχνά αναφέρεται ότι ο νόμος 1 του 2009 θα λύσει το πρόβλημα. Τι να γίνει εκεί. Ακόμα και ο πρόεδρος της Ρουμανίας κάλεσε το συνταγματικό δικαστήριο να εξετάσει τη συνταγματικότητα του νόμου. Είναι αλήθεια ότι το συνταγματικό δικαστήριο ε, ε, αποφάσισε ότι είναι συνταγματικό, αλλά τέσσερις δικαστές στο συνταγματικό δικαστήριο διαφοροποιήθηκαν. Δηλαδή γνωμοδότησαν διαφορετικά, λέγοντας ότι ο νόμος 1 του 2009 σαφώς απαλωτριώνει τους πρώην ιδιοκτήτες και είπε επίσης ότι ο νόμος δεν είναι συνταγματικός και ε, παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Ευχαριστώ. Η Μικαέλα Σαλαμούν. Θέλω να μιλήσω για το... Α, για το θέμα της επιστροφής ή αποζημίωσης στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Βέβαια, μια ε, ε, ξεκάθαρη νομική βάση θα ήταν καλύτερη και θα οδηγούσε σε ε, μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Όμως ακόμα η κωδικοποίηση αυτή είναι μακρά διαδικασία, συχνά πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι η διεθνής, διεθνής κοινότητα η τα διάφορα θεσμικά όργανα έχουν διάφορα μέσα στη διάθεσή τους για να αντιμετωπίσουν τα δικαιώματα ε, ιδιοκτησίας προσπαθώντας να επιτύχουν υψηλότερο βαθμό δικαιοσύνης στα συστήματα και τις διαδικασίες επιστροφών και αποζημιώσεων. Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρθηκε και αληθεύει ότι συχνά οι απαλωτριώσει στον, στο, στο, στο κομμουνισμό δεν είναι ε, θεμητέ λόγω ρατιών ετέμπορη, αλλά πολλέ φορέ πολλέ αποφάσει δείχνουν ότι η αντίληψη αυτή ε, έτυχε ευρεία ερμηνεία. Μπορεί δηλαδή να ήταν παραδεκτή απολωτρίωση αν υπήρχε κάποια σύνδεση με το παρόν ή με την ε, ε, κύρωση του πρωτοκόλου 1 της Σύμβασης. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μηχανισμούς Αναφέρομαι στη δήλωση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που είπε ότι αναφέρονται. Υπάρχουν, υπάρχει, υπάρχουν νομικές βάσεις που ήδη έχουν αξιοποιηθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ελάωρα Στέφαν. Uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα δώσω το λόγο στον συναδέλφό μου, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να μιλήσει συνοψίζοντας όλα τα σχόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Δύο μεθοδολογικά θέματα ερωτήθησαν από πλευρά των αξιωτήμων μελών του Κοινοβουλίου. Πρώτα απ' όλα, γιατί οι χώρε συμπεριλήφθησαν όπω συμπεριλήφθηκαν και γιατί δεν αναφερθήκαμε σε σχετικέ υποθέσει όπω την Ουγγαρία, Τσεχική Δημοκρατία. Η απάντηση είναι απλούστατη. Ε, αυτό ήταν, αυτή ήταν η σύμβαση. Έτσι τη διαμόρφωση το Ίδρυμα που μας ανέθεσε. Θα θέλαμε να αναφέρουμε τη Τσεχία και την Ουγγαρία. Είναι πολύ σχετικά. Ξέρουμε πώς πήγαν τα πράγματα. Εκεί δεν μπορούσαμε λόγω των όρων του συμβολέου. Ε, το θεωρούμε αυτό σαν ενθάρρυνση την πρότασή σας να επεκτείνουμε το πλαίσιο της μελέτης στο μέλλον τόσο ώστε να βοηθήσουμε τις χώρες που δεν έχουν καταλήξει σε κάποια απόφαση όπως είναι η Σερβία που ίσως θα θέλουν να εξετάσουν τα διάφορα μέσα όπως αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην Ουγγαρία, στη Τσεχική Δημοκρατία. Δεύτερον, η διαφθορά και το διοικητικό δηματικό εφαρμόζεται διάφορα μέτρα. Θα μπορούσαμε να είχαμε αναφερθεί ή αναφερθήκαμε σε αυτά, αναφερθήκαμε σε διάφορες χώρες, όμως είναι γενικά προβλήματα διοικητικής φύσεως και διαδικασιών λήψης αποφάσεων στις χώρες και ξεκινώντας να γράφουμε για διαφθορά και διοικητικό δυναμικό, δεν είναι κάτι που σχετίζεται μόνο με την ε, επιστροφή περιουσιών και μιλώντας για εφαρμοστικά, για προβλήματα εφαρμοσγής του νόμου υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την αποκατάσταση και τη μη αποκατάσταση περιουσιών που οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα. Ακίνητα, συμφωνίες για ακίνητα ε, που ακολουθήσουν και τις δύο πορείες. Είτε επιστραφούν είτε δεν επιστραφούν καταλήγει στα ίδια προβλήματα. Όμω, η έκθεση θα ήταν κάτι διαφορετικό αντί αυτή η περίπτωση. Η έκθεση για το δυναμικό των θεσμών σε αυτέ τι χώρε. και αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν μα ανετέθη να συγγράψουμε. Προσπαθήσαμε να τα κρατήσουμε όλα αυτά διαχειρίσιμα και να αναφερθούμε μόνο στην ιδιοκτησία, αλλά μα ανεθάρρυνε το ενδιαφέρον των που δημιούργησε η μελέτη και περισσότερα στοιχεία θα πρέπει να παραχθούν και θα πρέπει να γίνουν συγκρίσεις και με άλλες χώρες. Ίσως με η Πολωνία, η Τσεχική Δημοκρατία και η Ουγγαρία θα είναι χώρες οι οποίες θα μπορούσαν να αναφερθούν και αυτό θα ήταν πολύ επικοδομητικό. Ευχαριστώ πολύ. Από ό,τι κατάλαβε παρεμβάσει των συναδέλφων, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα υπάρχει και βούληση να παραμένει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Μεταξύ άλλων, οι πτυχέ που αναφέρθηκαν τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι απαντήσει που μόλι ακούσαμε ε, μα οθούν ε, Προ μια τέτοια αξιολόγηση ενδελεχέστερη επ' αυτού του θέματος. Θα ήταν λοιπόν κάθε απόφαση επί τη να την αφήσουμε για το μέλλον. Θα πρέπει η επικεφαλής των συντονιστών να αποφασίσει θα γίνει με την αναφορά που παραμένει ανοιχτή και θα μιλήσουμε συνεδρίες των συντονιστών για το θέμα. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε αντιστράψει, έχουμε, αναβάλει τη σειρά συζήτησης και έχουμε την έκθεση την για τη διερευνητική αποστολή στην Καμπανία. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στη συνάδελφο Μέρκης επικεφαλής, που είναι επικεφαλής αντιπροσωπείας της αποστολής αυτής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Την περασμένη εβδομάδα μεταβήκαμε στην Καμπανία για δυόμιση μέρες, επτά, άτομα είχε η αντισωπία, τρία, τρεις βουλευτές ε, του Ευρωκοινοβουλίου και τέσσερις από Ιταλικής πλευράς. Λάβαμε πάρα πολλές αναφορές σχετικά με το ζήτημα των αποβλήτων και τη μη εφαρμογή της οδηγίας για τα απόβλητα στην Καμπανία και ιδιαίτερα αυτές οι αναφορές γίνονταν δικά με τον ε, αποτεφρωτήρα και τις εκπομπές στην ε, Ατσέρα, στις ε, χωματερές, παράνομες χωματερές αλλά και ανοιχτούς χώρους ταφής Μεταβήκαμε λοιπόν επί τόπου για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα στον επόμενο και από εμπειρογνώμονες. Μπορώ να σας ε, αναφέρω κάποιες αρχικές εντυπώσεις διότι η έκθεση θα οδηγήσει σε κάποια συμπεράσματα αλλά περιμένουμε να είναι έτοιμη τον Ιούνιο. Λοιπόν, οι εντυπώσεις μας. Πρέπει να πω ότι οι αρχές έδειξαν ιδιαίτερη συνεργασία, επιθυμία για συνεργασία και πήγαμε σε διάφορες περιοχές. Πρόσφατα υπήρξαν ε, τοπικές εκλογές στην ε, Καμπανία σε ορισμένες επαρχίες και συζητήσαμε με τον πρόεδρο της περιφέρειας ο οποίος μόλις είχε διοριστεί δύο μέρες ακριβώς πριν να το συναντήσουμε. Ε, συνεργασία μας λοιπόν ήταν εξαιρετική. Την πρώτη μέρα είχαμε κάποιες ε, δυσκολίες και σε ό,τι φορά την πρόσβαση με τους ε, αναφέροντες και με τον τύπο. Αλλά αυτό ρυθμίστηκε γρήγορα ο τύπος δεν είχε τη δυνατότητα να προσέλθει και προς τις περιοχές που επισκεφθήκαμε και είπαμε ότι η διαφάνεια δεν υπήρχε ούτε για, τον, ούτε για τον τύπο ούτε για, την, για τους ε, αναφέροντες και αν αυτό συνεχιστεί θα αποχωρήσουμε. Οι αρχές λοιπόν έδειξαν ιδιαίτερη συνεργασία και την επόμενη μέρα δόθηκε άδεια στους δημοσιογράφους αλλά και στις, ε, σε τοπικές αρχές που δεν είχαμε μέχρι τούδε ποτέ πρόσβαση αλλά και τους αναφέροντες. Ε, μόλις ρυθμίστηκε αυτό το ζήτημα θα ήθελα να πω ότι οι εντυπώσεις μας ε, ήταν ότι λόγω της πολιτικής αλλαγής που είχε γίνει μετά από τις τοπικές εκλογές και η νέα, η νέα αρχή, οι νέοι αιρετοί άρχοντες ε, πιστεύουμε πως ε, θα φέρουν τις απαραίτητες αλλαγές και την εφαρμογή των, ε, της κοινωτικής νομοθεσίας. Αυτό ενδέχεται να αποτελέσει την απαρχή ενός διαλόγου με τις τοπικές αρχές της Καμπανίας και τους πολίτες, κάτι το οποίο ε, απουσίαζε μέχρι τώρα. Αυτά λοιπόν τα θέλαμε να σας πούμε. Μεταξύ αυτών ε, είδαμε πως υπήρξε απουσία ενός επικοδομητικού διαλόγου ανάμεσα στους αναφέροντες ε, και τις αρχές ε, και διαπιστώσαμε, πώς δεν το πω, πως ο διάλογος ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα και αυτός δύναται να βελτιωθεί περαιτέρω. Είπα πως υπάρχει ελπίδα για μια νέα αρχή μετά από τις αλλαγές στην περιφέρεια. Τι συνέβη. Εμείς επισκεφθήκαμε ε, χωματερές, των ε, ε, ανοιχτές, τοποθεσίες ε, για την απόρριψη αποβλήτων και θα έλεγα ότι Όντως υπήρξε, υπήρχε μάλλον έλλειψη διαλόγου και διαφάνειας. Ευτυχώς ε, μπορώ να πω ότι η υποστολή μας ε, επέφερε κάποιες αλλαγές. Λόγω του ότι φτάσαμε εκεί, πήγαμε εκεί, ξεκίνησε ένας νέος διάλογος, υπήρξε δυνατότητα πρόσβασης από πλευράς πολλών ε, το τοπικών αρχόντων στις περιοχές αυτές, στις κομματερές, στις χιτά κλπ. Τώρα, οι οδηγίες αυτές περί αποβλήτων, ε, οι αρχές γνωρίζουν ότι μπορούν να εφαρμοστούν και αυτό τελεί απέτηση τόσο των αρχών όσο και των ε, πολιτών. Μας δόθηκε η εντύπωση πως δεν υπάρχει ένας ολοκληρωμένος κύκλος διαχείρισης αποβλήτως στην καμπανία. Φυσικά σα λέω κάτι το οποίο έχει ήδη υποθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μέσω μιας απόφασης αυτής τη 4 Μαρτίου 2010 που ορίζει ότι η Ιταλία δεν συμμορφώνεται με, με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτή η έλλειψη λοιπόν κύκλο διαχείρισης των αποβλήτων οδηγεί στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η καμπανία που αφορά τις χωματερές αλλά και, τις, ε, και τους τα μηχανήματα κάψης, ε, τις εγκαταστάσεις κάψης των αποβλήτων. Ε, επισκεφθήκα το Εθνικό Πάρκο του Βεζούβιου που όπως ε, γνωρίζετε είναι μεταξύ των μνημείων που έχουν ενταχθεί στην UNESCO και στην περιοχή υπάρχουν ε, απόβλητα τα οποία απορρίπτονται και ελπίζω και οι αρχές ε, να το ρυθμίσουν το ζήτημα. Μια άλλη τοποθεσία θεωρείται πως ε, και αυτή θα εγκαταληφθεί και θα πάψει να χρησιμοποιείται. Η τρίτη εντύπωση είναι πως ε, η διαφάνεια μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω, εάν ε, δεν παρέχεται δυνατότητα πρόσβαση στους πολίτες, στις τοπικές αρχές, ούτε στους, ε, στον τύπο, τα στοιχεία δεν μπορούν να επαληθευτούν. Και θεωρώ πως εάν δεν υπάρχει διαφάνεια τότε δεν μπορούμε να έχουμε και τον απαιτούμενο διάλογο και ζούμε σε ένα κλίμα έλλειψης εμπιστοσύνης, δυσπιστίας. Υπήρξαν λοιπόν κάποια θετικά μηνύματα, όχι μόνο σε ό,τι φορά την συνεργασία των τοπικών αρχών και των εμπειρογνωμών και των αναφερόντων, αλλά όλα αυτά πραγματικά τα διαπίστωσαν και οι Ιταλοί συνάδελφοι. Πρόκειται ένα, τα απόβλητα είναι ένα ζήτημα εγκάρσιο. Το ζήτημα των απόβλητων πολιτικοποιήθηκε στην ε, Καμπανία και το ένα κόμμα επέριπτε στο άλλο είναι επαναλαμβάνω ένα εγκάρσιο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει όλα τα κόμματα και όλους τους πολίτες. Θα ήθελα να καταλήξω λοιπόν με, αυτό, με αυτή την αχτίδα ελπίδας. Ευχαριστώ την συνάδελφο Μέρκελ. Αν επιθυμεί κάποιος να λάβει το λόγο, ο συνάδελφος Γιάρ. <coughs> Äh, λοιπόν, θα ήθελα να προβώ ένα μικρό σχόλιο για να συμπληρώσω αυτό που είπε ο κεφαλής αντιπροσωπείας. Πράγματι σωστά τα είπε, όσα είπε. Ήταν ένα ταξίδι εντυπωσιακό για όλους τους ε, συμμετέχοντες και η Επιτροπή Αναφορών μπόρεσε να δει επιτόπου τα όσα συνέβαιναν με αυτά τα απόβλητα και μπόρεσε να, μπόρεσε να αντιληφθεί καλύτερα την κατάσταση. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η επίσκεψη διότι μπορέσαμε να συνοδεύσουμε συνοδέλφους ε, ήταν μια επίσκεψη μη επίσημη αλλά θέλω να συμπληρώσω αυτό που είπε η επικεφαλής αντιπροσωπείας δηλαδή ότι ε, υπήρχε αυτό το πρόβλημα λοιπόν σχηματίσαμε μια εικόνα και θεωρήσα ότι αυτές οι χωματερές ήταν κάτι προσωρινό. Αλλά διαπιστώσαμε ότι το προσωρινό του πράγματος ε, κράτησε πολύ και κρατάει. Έχω την εντύπωση ότι βασιστήκαμε πολύ σε τέτοια παρεμφερή συστήματα και προσωρινές λύσεις. Και αυτό είναι πρόβλημα. Και νομίζω ότι θα προκύψει εκ νέου το πρόβλημα θα εξαντληθούν οι, οι, οι φυστάμενες χωματερές, δεν θα μπορούν να δεχτούν άλλα απόβλητα και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια νέα λύση. Χρειαζόμαστε περισσότερο διάλογο, μεγαλύτερη διαφάνεια και πάνω απ' όλα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε τον διαχωρισμό των αποβλήτων και πιστεύω ότι ήταν επιτυχία τελικά αυτή η επίσκεψη. Γιατί σχηματίσαμε εικόνα, όπω σα είπα. Και στην τελευταία μέρα, αφού μιλήσαμε με τι τοπικέ αρχέ, εκπροσώπου τοπική αυτοδιοίκηση, είδαμε ότι το έργο του είναι δύσκολο. Πρέπει να πάρουν αποφάσει επιτόπου διάφοροι αρμόδιοι. Και είναι αισθητά τα αποτελέσματα μια αποφάσεως πολιτικής για τα απόβλητα. Από πρώτο χέρι οι κάτοικοι αντιλαμβάνονται αν είναι λάθος ή σωστή μια απόφαση για τα απόβλητα. Ήταν υπέροχο βέβαια που οι αναφέροντες ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι που πήγαμε σαν αντιπροσωπεία όμως δεν πρέπει να τους ε, διαψεύσουμε τις ελπίδες τους θα πρέπει να γίνουν σοβαρέ συνομιλίε και θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε λύσει οι οποίε θα μπορούν να είναι εφικτέ, εφαρμόσιμε. Ευχαριστώ, Γιώργαν. E θα ήθελα να υπενθυμίσω, συνάδελφοι, τον λόγο για τον οποίο μετέβημε στην καμπανία. Οι αναφορές αφορούσαν τον, τις, ε, τον, την αποτέφρωση αλλά και τις, ε, τις ταφές ε, των, ε, της χωματέρας συγγνώμη σε ό,τι φορά τον αποτεφρωτήρα όλοι διαπιστώσαμε πως μιλάμε για μια κατάσταση υψηλότερης τεχνολογίας και που δίνει ένα καλό αποτέλεσμα ιδίως από πλευράς περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά κάποιες διευκρινήσεις θα ήθελα να κάνω προς την Αλφα Μέρκενς ε, κοιτάξτε, συνάδελφε, οι χωματερές στην Καμπανία με κρατικό νόμο ε, θεσπίστηκαν ως χώροι εθνικού ενδιαφέροντος και έτσι δεν μπορούν οποιοδήποτε ούτε καν οι δήμαρχοι να επισκεφθούν τον χώρο. Εάν ε, θεωρεί και μάλλον αυτό το διάταγμα θεωρήθηκε απαραίτητο διότι οι επιτροπές ήταν τόσο πολύ άριθμες και δεν μιλάμε για εκατοντάδες άτομα τα οποία είχαμε τη δυνατότητα να συναντήσουμε εμείς, αλλά μιλάμε για χιλιάδες άτομα τα οποία εμπόδιζαν, παρεμπόδιζαν την πρόσβαση στις ε, χωματερές. Ως εκ τούτου η κυβέρνηση βρέθηκε στην κατάσταση να χρειαστεί να ε, αποφασίσει πως πρόκειται για έναν χώρο εθνικού ε, ενδιαφέροντος και τον έθεσε υπό την προστασία του στρατού. Και εσείς στην Βόρεια Ευρώπη που εκπλήσεστε με την παρουσία του στρατού εκεί, αλλά ε, για μας τους Ιταλούς όταν βλέπουμε τον ένστολο, το στρατιώτη, αυτό μας καθησυχάζει. Όχι όπως συμβαίνει στην Ανατολική Ευρώπη, εμείς λοιπόν εμάς μας καθησυχάζει ο ένστολος και θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό το οποίο επιτηρούν και εποπτεύουν ε, είναι ασφαλές. Φυσικά η του Γκαγιάνο μαζί μας είχα τη δυνατότητα να διαπιστώσετε πως είναι ένας χώρος ασφαλής. Κανείς δεν θέλει να αποκρύψει στην Ευρώπη, στον κόσμο ότι πρόκειται για μια χωματερή που βρίσκεται στην περιαστική περιοχή. Φυσικά υπάρχουν κάποια προβλήματα στην, ε, στο Τερζίνιο. Οι τοπικές αρχές μας διασφάλισαν ότι η άλλη χωματερή που που φέρει το όνομα Βιτήλο δεν ε, πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, δεν πρόκειται να ανοίξει προς χρήση και ουσιαστικά χωματερές προσωρινού χαρακτήρα δεν υπάρχουν. Μια χωματερή παραμένει πάντα χωματερή και θα πρέπει να ε, τύχει ε, σωστή διαχείριση και να κλείσει. Εμείς ε, που είμαστε από την καμπανία επιθυμούμε να μην υπάρξουν νέες χωματερές για να συμβεί κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε νέες εγκαταστάσεις αποτέφρωσης. Χρειάζεται να υπάρξει μια διαφοροποιημένη συλλογή των απορριμμάτων και για να συμβεί κάτι τέτοιο μας χρειάζεται χρόνος και πόροι. Ας ε, κοιτάξουμε ως Ευρωπαϊκό Θεσμικό Όργανο και την πηγή των πόρων των οικονομικών, διότι σε μια περίοδο διαδομένης κρίσης τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίω, εκεί όπου δεν υπάρχουν πόροι, καταστάσεις και διατάγματα ε, βελτιωτικά δεν μπορούν να υπάρξουν ε, ούτε εξηγένση θέσεων. Ο Μπελίν, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την επικεφαλής της αντιπροσωπείας ε, Μέρκελ και όλους όσοι έλαβαν μέρος σε αυτήν την αποστολή και, την, και τον γραμματέα αλλού. Εγώ δεν είμαι μόνο ευρωβουλευτής, αλλά είμαι Ναπολιτάνος ε, και είμαι υπερήφανος ε, που γεννήθηκα στην περιοχή. Η επίσκεψή μας ήταν μια στιγμή υψηλής ε, δημοκρατίας, υψηλού δημοκρατικού χαρακτήρα. Υπήρχε δυνατότητα και να μπορέσετε και εσείς κύριοι βουλευτές να δείτε μια τραγική κατάσταση, αλλά μια εξαιρετική περιοχή που ήταν και η πατρίδα της ε, Μάγνια Γκρέτσια ήταν η πρωτεύουσα της ε, περιοχής. Δεν πρέπει λοιπόν να στροφοκαμιλίζουμε. Ε, μεγάλη δυσκολία αντιμετωπίσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες ε, αυτές οι εικόνες της πόλης της Νάπολης καλυμμένης από σκουπίδια είναι δύσκολο να την καταπιούμε και να την ξεχάσουμε αλλά τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει βελτίωση, αναφίβολα. Ε, οι χωματερές ε, δημιουργήθηκαν διότι υπήρχε ένα κατεπήγον ζήτημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί, αλλά εμείς στη συνεργασία με τους τεχνικούς και τις ε, αρχές διαπιστώσαμε πως έχει αναλυφθεί μια πρωτοβουλία όχι μόνο σε ρεφορά την διαφοροποιημένη επιλεκτική διαλογή των σκουπιδιών διότι το 5% θα πετύχουμε το, ένα ποσοστό της τάξης του 50% μέσα στο επόμενο έτος, ε, κάτι το οποίο είναι κάτι που μας ανακουφίζει, όπως και η διαχείριση του συνολικού κύκλου των απορριμμάτων είναι ένα γεγονός. Ε, Στη συνάντηση που είχαμε με τους εκπροσώπους των περιφερειών, ακούσαμε για ένα πρόγραμμα σχετικά με τη μείωση των ε, απορριμμάτων, όχι μόνο για τον ολοκληρωμένο κύκλο διαχείρισης των απορριμμάτων. Υπάρχει λοιπόν ελπίδα. Θεωρώ ότι με βάση αυτή την επίσκεψη θα πρέπει να ε, να ταινίσουμε μια αισιοδοξία το μέλλον. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε στους πολίτες της ε, καμπανίας αυτά που υποσχεθήκαμε κατά την επισκεψή μας. Υποσχεθήκαμε ότι μέσα σε ένα χρόνο η, Επιτροπή, η, συγγνώμη, η Επιτροπή της Επιτροπής Αναφορών θα επιστρέψει και θα ε, ε, επιβεβαιώσει τις ε, προόδους που έχουν επιτευχθεί. Υπενθυμίσαμε στους τοπικές αρχές ε, που είναι και αρχές οι οποίες ε, προ ο, λίγων μηνών ανέλαβαν το να εκτελέσουν το έργο τους ε, διότι είναι πρόσφατα εκλεγμένοι ότι η Ευρώπη δεν θα ξεχάσει αυτή την γη και επαναλαμβάνω πως θεωρώ ότι η επίσκεψή μας αποτέλεσε μια σημαντική δημοκρατική στιγμή ευχαριστώντας ε, και τον πρόεδρο Ματσόνη την πρόεδρο μάλλον Ματσόνη της Επιτροπής μας ε, που έθιξε σε το ζήτημα της καμπανίας ε, στην Επιτροπή μας και μπόρεσαν όλοι να διπιστώσουν ότι οι κάτοικοι της περιοχής ότι η Ευρώπη δεν βρίσκεται μακριά. Όταν ε, της ε, ζητείτε κάτι, δρά, μεταβαίνει επί τόπου. το γεγονός ότι υπάρχουν τόσοι ε, πολίτες που δεν προσφέρουν στις κάλπες κατά των ε, ε, ευρωεκλογών οφείλεται σε μια ιδέα που έχουν εσφαλμένα δημιουργήσει οι πολίτες και να ευχηθούμε ότι στο εγγύς μέλλον με έξοδα των βουλευτών, όχι με έξοδα του Κοινοβουλίου, να επιστρέψουμε στην περιοχή για να γνωρίσουμε τις ομορφιές αυτή τη γη και όχι να ασχοληθούμε με έκτακτα γεγονότα. Δεν υπάρχει κανείς άλλος που να έχει ζητήσει το λόγο. Ε, διευκρινίζω ότι αυτή είναι μια πρώτη φάση συζητήσεων σχετικά με την αποστολή στην ε, καμπανία. Μετά θα περάσουμε στην πρόταση, μάλλον στην αναφορά από τον επικεφαλής της Ελληνικής στην Επιτροπή μας και Όπω είπε η κυρία Μέρκε, αυτό θα στα, χέρια μας το έγγραφο μέχρι τον Ιούνιο. Η κυρία Μέρκε. υπενθύμησε πως ο Πρόεδρο τη Επιτροπή Καμπανίας που συναντήσαμε είχε μόλις αναλάβει καθήκοντα και με την ευκαιρία αυτή ως πρόεδρος της Επιτροπής αλλά και με τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής κάλεσα τον πρόεδρο της ε, Περιφέρειας και με τον σύμβουλο ο οποίος θα διοριστεί στο εγγύς μέλλον ελπίζουμε και για θέματα διαχείρισης αποβλήτων να έρθουν εδώ στις Βρυξέλλες στην Επιτροπή μας και να μας μιλήσουν για τις λεπτομέρειες που δεν μπόρεσαν να μας παράσχουν προ την περσμένη εβδομάδα διότι είχε λάβει καθήκοντα επαναλαμβάνω μόλις πριν από δύο μέρες και για μια διευκρίνηση συναντήσαμε κάποιες δυσκολίες και συμφωνώ με την συνάδελφο Μέρικης ότι δεν ήταν ευχάριστες οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε κατά την επίσκεψή μας, αλλά το ότι χρειάστηκε να αναθέσουμε τη διαχείριση κάποιων ε, περιοχών, κάποιων χωματερών ε, στην, υπό την προστασία του στρατού καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα ζήτημα πολύ σοβαρό την πρώτη μέρα λοιπόν ε, βρήκαμε απέναντι μας ένα τείχο διότι δεν είχαμε επισημοποιήσει την δυνατότητα πρόσβασης στους χώρους ε, ε, αυτούς και την προσεχή ημέρα όμως ε, λάβαμε αυτές τις άδειες, υποβάλαμε το αίτημά μας, λάβαμε λοιπόν την άδεια για την επίσκεψη και τόσοι πολίτες όσο και ο τύπος που ήταν παρόν είδε πως ε, η πρόσβαση είναι δυνατόν ε, να επιτευχθεί αρκεί να διατηρηθούν οι διαδικασίες οι οποίες επιβάλλονται λόγω της καταστάσεως που επικρατεί σε, αυτές τις, ε, σε αυτούς τους χώρους, σε αυτές τις εγκαταστάσεις και κάτι ακόμα ε, η κατάσταση είναι τραγική, γι' αυτό είναι γεγονό. Μιλάω για την κατάσταση η οποία αποκρισταλώθηκε στην απόφαση της 4 η Μαρτίου. Απόφαση του δικαστηρίου που αναφέρεται στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Καμπανία και κατεγγέλθηκαν στις αναφορές μέχρι τον Ιούλιο του 2007. Αυτή η απόφαση του δικαστηρίου αναφέρεται στην κατάσταση που κρατούσε τον Ιούλιο 2007. Από τότε ε, ξεκίνησε μια διαδικασία πέραν του δράματος λοιπόν το οποίο δεν μπορέσαμε να διαπιστώσουμε αλλά βέστος υπάρχει μια κατάσταση αρέσκειας εμείς χρειάστηκε να, να δούμε αν τα τελευταία δυόμιση χρόνια κάτι έχει συμβεί εάν έγιναν κάποιες παρεμβάσεις προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση και αυτό είναι κάτι το οποίο θα συμπεριληφθεί στην έκθεση, αλλά σίγουρα τα πράγματα ε, προχώρησαν, κουνήθηκαν ε, λίγο. Ε, φυσικά υπάρχουν οι ανησυχίες των πολιτών σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για το περιβάλλον, οδηγία για την απόβλητα και για την υγεία. Αυτό θα το ελέγξουμε μετά από τα τόσα στοιχεία που συλλέξαμε και από την τεκμηρίωση θα πρέπει να ξεκινήσουν πάντως ε, από την συνεργασία που έδειξαν οι αρχές και κάτι που τόνισε η κυρία Μέρκετς. Ε, θα εξετάσουμε λοιπόν εκ νέου το ζήτημα μου. Ο κ. Κοτσολίνο Νέφη, παρακαλώ, για το λόγο. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Έφτασα μόλις τώρα. Πιστεύω ότι αυτά που άκουγα που έλεγε η Πρόεδρος ε, αντικατοπτίζουν και τη δική μου προσωπική άποψη. Η κατάσταση που αντιμετώπισα εκεί θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολη, αλλά ξεκίνησαν και κάποιες προσπάθειες που πρέπει να ενθαρρυνθεί και να οδηγηθεί στο τέρμα. Έχουμε μία πρόκληση, μία σημαντική περιοχή της Νότιας ε, Ιταλίας να αποκτήσει τελικά ένα σύστημα ολοκληρωμένο συλλογής ε, και αποκομιδή των διαφόρων αποβλήτων, των αστικών και των βιομηχανικών. Έχουμε στην πλάτη μας πολύ δύσκολη κατάσταση, περίπλοκη, ε, που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια. Έγιναν προσπάθεια, γίνονται προσπάθειες τώρα και οι τοπικές αρχές κινούνται πάνω σε αυτό το δρόμο, σε αυτή την προσπάθεια. Είναι τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλονται και πιστεύω ότι η Ευρώπη θα πρέπει να μπορεί να συνοδεύσει όλη αυτή την προσπάθεια να παρακολουθεί με προσοχή την προσπάθεια, να την υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια και πάνω απ' όλα να επαγρυπνεί διότι τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν τους επόμενους μήνες ε, να μην γίνει ε, τέτοια που να μας οδηγήσουν στην ίδια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ε, και τελικά πρέπει να αντλήσουμε μαθήματα από την έκτακτη ανάγκη, το άνοιγμα χωματερών, ε, και εκεί που θα έπρεπε να προστατευτεί η κληρονομιά το, η περιβαλλοντική της περιοχής να προστατευτεί ή να, έχουμε, ε, να μην έχουμε εγκαταστάσεις που είναι απειρχιωμένες για την επεξεργασία των αποβλήτων. Ε, γίνεται η μάχη, πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή τη μάχη που έχει δρομολογηθεί επί δύο σημείων που θεωρώ ότι είναι θεμελιώδη σημασία. Από τη μία πλευρά θα πρέπει να μειωθεί η παραγωγή των αποβλήτων, αυτή είναι η πραγματική πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι πλευρά νοοτροπία και συμπεριφορά των πολιτών και θα πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα περισυλλογή και κατεργασίας των αποβλήτων πιο προχωρημένο πλευράς οικολογικής και να γίνει και σωστή διαφοροποίηση των αποβλήτων. Και θα πρέπει να συμμετάσχει και η τοπική κοινότητα, η τοπική αυτοδίκηση στην όλη προσπάθεια. Διεφάνει και κάτι και είναι αποτέλεσμα μεγάλης εμπειρίας το μεγάλο πρόβλημα επικοινωνίας και σχέσεων με τους πολίτες. Θα πρέπει και από αυτή την έποψη να συμβάλλουμε. Ε, διότι και στις πιο δύσκολες καταστάσεις και στις καταστάσεις κατεπίγουσες, άκρως κατεπίγουσες όπου κινδυνεύει η υγεία των πολιτών, πρέπει να υπάρχει ε, μια διαφάνεια και μια δημοκρατική συμμετοχή όσον αφορά τα όσα κάνει η δημόσια διοίκηση. Γι' αυτό είναι σημαντική η παρουσία μας και η αποστολή μα και θα είναι και σημαντικό να επιστρέψουμε με μια νέα αποστολή και σε ένα ενάμιση χρόνο για να δούμε και κατά πόσο ε, υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών και τη τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι προαπαιτούμενο για την επίτευξη των στόχων που έχουμε προτείνει ε, που κατά κάποιο τρόπο πιστεύω ε, ήταν και η εικόνα που σχημάτισε η αποστολή αυτή ε, τις τέσσερις μέρες που μείναμε στην καμπανία. Ευχαριστώ, συγγνώμη καθυστέρηση, ευχαριστώ κύριε Κοτσολίνο. Δεν ξέρω θέλει να μιλήσει ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Μάρκ Λεμέρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά το θέμα αυτό, νομίζω ότι είπατε τα ουσιώδη σχετικά με την ε, έκθεση. Εγώ δεν έχω πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. Η απόφαση ελήφθη από το δικαστήριο στις 4 Μαρτίου του 2010, όπως μας είπατε. Σε αυτή την υπόθεση και σε αυτή την περίπτωση στέλνουμε επιστολή προς το κράτος μέλος για να ρωτήσουμε ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για να συμμορφωθεί με το κοινοτικό δίκαιο. Αυτό κάναμε όσον αφορά την Ιταλία και αναμένουμε την απάντηση η οποία θα πρέπει να δοθεί το δίμηνο μετά την αποστολή της επιστολής όπου η Ιταλία θα μας δείξει πώς θέλει να χρησιμοποιήσει το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ποια μέτρα ελήφθησαν. Να υπενθυμίσω κάτι στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας για την εκτέλεση των αποφάσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί μια επιταχυμένη διαδικασία διότι εδώ στείλαμε μια προειδοποίηση όσον αφορά την εκτέλεση του άρθρου 260 ε, εδώ βρισκόμαστε όσον αφορά την παρακολούθηση εκτελέσεως της αποφάσεως αυτής που έχει ληφθεί. Σας ευχαριστώ. Κύριε εκπρόσωπε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορούμε να ολοκληρώσουμε και αυτό το σημείο τη ημερήσια διάταξη. Επόμενη συνάντηση, μπορούμε να ενωθούμε. Πάμε. Στο επόμενο σημείο της ημερήσια διάταξη, το 16, διότι το 15 ε, ανεβλήθη όπως συμφωνήσαμε για άλλη συνεδρίαση κατόπιν συμφώνου γνώμης των συντονιστών των ομάδων το σημείο 16 είναι αναφορά 265 του 2007 της Νατάλια Γκονζάλες Μενέντες που δεν είναι παρούσα. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αντρέ Κόμπε, να αναφερθεί στο θέμα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, για λόγους συντομίας, θα ήθελα να πω ότι τα σημεία 16 ως 20 ασχολούνται με την ανοσφαιρική ρήπανση και τα αιωρούμενα σωματίδια και πώς αντιμετωπίζουν το πρόβλημα τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άμα επιτρέπετε λοιπόν θα ήθελα σύντομα να εξηγήσω την όλη διαδικασία, ε, την τοποθέτηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά να αναφερθώ σε μια δήλωση όταν θα διατρέξω τις διάφορες αναφορές σχετικές με το ζήτημα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με τη διαδικασία. Συμφωνείτε, συμφωνείτε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όσον αφορά τα αιωρούμενα σωματίδια, η ουριακή τιμή ίσχυε από το 2005 και αυτό επιβεβαιώθηκε και από τη νέα οδηγία που υιοθετήθηκε το 2008, η οποία όμως επιτρέπει υπό κάποιες συνθήκες τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να έχουν χρόνο στη διάθεσή τους μέχρι τις 2011 για να συμμορφωθούν ε, με τις οριακές τιμές όσον αφορά το, τα αιωρούμενα σωματίδια, το PM10, 350.000 άνθρωποι κάθε χρόνο πεθαίνουν πρώιμα από την ατμοσφαιρική ρήπανση, κυρίως λόγω των αιρούμενων σωματιδίων, το PM10 όπως αποκαλείται, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το λόγο έχει αναλάβει την υποχρέωση να εφαρμόσει την οριακή αυτή τιμή και να κινηθεί σοβαρά για την εφαρμογή αυτή. Και σχετικά με αυτό θέλω να πω ότι διάφορα διαδικασίες παράβασης έχουν ήδη δρομολογηθεί. Ε, είναι σε διαφορετικές ε, φάσεις εκτελέσεως διότι με αυτή τη συμπληρωματική διάταξη που επιτρέπει ε, περαιτέρω χρονικό διάστημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί και αποτιμά ε, συγκεκριμένες κοινοποίησεις σχετικά με τα κάτι μέλη που χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Σχετικά με αυτό θα μπω σε λεπτομέρειε, θα αναφερθώ σε συγκεκριμένε οδηγίε και θα αναφέρομαι πώ πήγαν τα πράγματα σε συγκεκριμένε υποθέσει. Τώρα, όσον αφορά την αναφορά 265, ε, μιλάμε για υπερβολική έκθεση σε ατμοσφαιρική ρήπανση, κυρίως σκόνη και θόρυβο. Υπάρχει χαλιβουργείο ε, στο Κιχόν ε, θα πρέπει να δούμε ότι και το 2008 υπάρχει και πάλι υπέρβαση των οριακών τιμών για τα σωματίδια, το PM10, στην περιοχή. Δεν έχει δοθεί παράταση, δεν έχει ζητηθεί παράταση χρονική. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία παράβασης ε, προκαιρού και τώρα στις 22 Μαρτίου εκδώσαμε αιτιολογημένη γνώμη κατά της Ισπανίας ε, για την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου όσον αφορά τα αερούμενα σωματίδια, το PM10 Περιμένουμε λοιπόν μια απάντηση από τον λόγο κάτω μέλος για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Το Κιχόν είναι μια περιοχή με υπερβάσεις, οπότε θα ε, κάνουμε την αξιολόγηση ανάλογα με την ε, ε, κατάσταση που κρατεί. Λόγω λοιπόν της ιδιαιτερότητας της κατάστασης, λόγω τοπικής υπέρβασης κοντά στο Χαλιβουργείο, έχουν άδεια για IPPC, Πώς όμως αυτό επηρεάζει την ποιότητα του τροσφαιρικού αέρα ε, είναι το θέμα. Κοντά στην ε, μονάδα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αξιολογηθεί περαιτέρω. Το πρόβλημα δεν έχει επιλύθει ακόμα, όπως προανέφερα, όσον αφορά το θόρυβο. Ο χάρτης θορύβου για το κηγόν ε, δόθηκε, έλειπαν οι χάρτες στην πρώτη υποβολή των στοιχείων από την Ισπανία, παρεσκέθησαν τώρα οι χάρτες, ζητήθηκαν σχέδια δράσεως που συσχετίζουν τα προβλήματα τα εντοπιστέντα μέσω των χαρτών θορύβου με συγκεκριμένα μέτρα διορθώσεως του προβλήματος και όλα αυτά αξιολογούνται, αναλύονται. Όμως η καταδική ανάλυση καταδεικνύει ότι το σχέδιο δράσης για το Κιχόν δεν έχει υποβληθεί. Και αν περί αυτού πρόκειται, θα ακολουθήσουμε και άλλη δράση, τόσο ώστε το σχέδιο δράσης τελικά να υπάρξει και να υποβληθεί. Αυτά όσον αφορά την αναφορά υπαριθμών 265. Ίσως θα μπορούσατε να προχωρήσετε και με το επόμενο, με το επόμενο σημείο. Αν μου λέτε ότι πάντα εσείς θα παίρνετε το λόγο, διότι εσάς έχω πάντα ως εκπρόσωπο της Επιτροπής όσον αφορά τα συναφή θέματα. Να αναφέρετε και τα άλλα και έτσι θα μπορέσουμε να εξετάσουμε και τις αναφορές μαζί και τι δύο. Καλώς λέει ο κόσμο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την αναφορά 831 Έχουμε υπέρβαση ερωμένων σωματιδίων ΑΣ10 κοντά σε εγκατάσταση, σε μονάδα βιομηχανική. Εδώ η μονάδα αυτή δεν καλύπτεται από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όμως η κατάσταση εδώ διαφέρει. Επετεύθη η μόρφωση με τα όρια το 2008 και πιστεύουμε ότι τώρα δεν υπάρχει εντοπισμένη παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας όσον αφορά τη βιότα του σφαιρικού αέρα, όμως εντωμεταξύ είχαμε ανταλλαγές απόψεων με την ισπανική κυβέρνηση για να είμαστε σίγουροι ότι γίνεται σωστή αξιολόγηση στην περιοχή του ατμοσφαιρικού αέρα, διότι όπως σωστά λένε οι αναφέροντες, στη μονάδα μέτρησης έχει μετρηθεί η υπέρβαση, δεν είχε όμως ε, η υπέρβαση κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως σύμφωνα με τη σχετική διάταξη θα πρέπει στην, στην περιφέρεια να διαπιστώσουν κατά πόσο η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Και θα μας ενημερώσουν οι αρχέ Αρχές ε, σχετικά με την κατάσταση του ατμοσφαιρικού αέρα. Τώρα, όσον αφορά την επόμενη αναφορά, Θα πάω στο σημείο 18. Είναι η αναφορά 1459 του 2007 όσον αφορά τη βιομηχανική ρήπανση Συγγνώμη, λέει Πρόεδρος, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, να εξετάσουμε τις δύο αναφορές μαζί, διότι είχαν ανατεθεί στον ίδιο συνάδελφο και αφορούν το ίδιο θέμα. Θα διακόψουμε, θα ζητήσω από συναδέλφους να θέλουν να μιλήσουν και μετά θα περάσουμε στο σημείο 18, το οποίο έχετε αναλάβει εσείς, έχετε αναλάβει εσείς αυτή την αναφορά. Μάιερ, συνάδελφος Μάιερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λαμβάνω το λόγο μόνο και μόνο για να πω πως οι αναφορές 15, 16 και 17 ζητώ να παραμείνουν ανοιχτές διότι οι 16 σύμφωνα με την Κομισιόν υπάρχουν, υπάρχει εκκρεμότητα, δηλαδή αναμένεται η απόβονηση της Ισπανικής Κυβέρνησης και οι 17 Επίσης, διότι οι αναλύσεις που έγιναν σχετικά με, τον, με την πόλη Αλκανής απαιτεί μια περαιτέρω εμβάθυνση από πλευρά Κομισιόν. Παρακαλώ λοιπόν πρόεδρε να παραμείνουν ανοιχτές οι δύο αυτές αναφορές. Η συνάλληψη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφέρω σχετικά με την παριθμόν 16 αναφορά αυτή την οποία αναφέρθηκε και η Κομισιόν ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μου θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες επαναλαμβάνω υπάρχουν μια σειρά διορθωτικών μέτρων τα οποία ελήφθησαν και εφαρμόζονται σε σχέση με την ηχορύπανση που θα καταστούν ε, ε, λειτουργικά από τον Ιούνιο του 2010. Θα, λοιπόν, να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, αλλά μόλις όλοι οι μηχανισμοί τεθούν σε λειτουργία κάτι το οποίο έχει επιβάλει η τοπική κυβέρνηση στην ε, επιχείρηση. Η επιχείρηση λοιπόν θα έχει κάποιο, έχει κάποιο χρόνο στη διάθεσή της για να συμμορφωθεί και τον Ιούνιο 2010 θα πρέπει να έχουμε νέα στοιχεία. Τώρα σε ό,τι φορά την ποιότητα του αέρα που είναι η άλλη πτυχή της αναφοράς ε, η Κομισιόν αναφέρει τη στοιχεία του 2008 αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες μου τους, τα τρία τελευταία χρόνια υπήρξε μια σημαντική μείωση των επιπέδων ρήπανσης όσο σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ημερών κατά τον οποίο υπερβαίνεται ο, η, οριακή τιμή το ΑΕΣ 10 δεν ξεπέρασε για καμία μέρα τον το ανώτατο αυτό όριο τιμής. Ε, τα δύο τελευταία λοιπόν χρόνια αυτό το ανώτατο μόνο μία φορά το υπερεύει η ρήπανση. Δεν ξέρω λοιπόν αν η Κομισιόν έχει στα χέρια της αυτόν το στρατηγικό χάρτη για την ε, ηχορύπανση, αλλά τα στοιχεία που έχω εγώ δεν συμπίπτουν με τα σχόλια της Κομισιόν. Θα ήθελα λοιπόν να γίνει κάποια διευκρίνηση. Η Κομισιόν. Δεν ci sono altri interventi. Η Κομισιόν έχει το λόγο. Τι να κάνω, Πρόεδρε. Η πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο. Μία σύντομη παρέμβαση, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα θέλω να πω ότι και εγώ είμαι υπέρ να παραμείνουν ανοιχτές οι αναφορές που έχουμε ενώπιον μας σήμερα. Ελπίζω η Κομισιόν να παρακολουθήσει τις εξελίξεις τους δύο αυτούς φακέλους και να λάβει τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες το, 17 αναφέρονται, στις 17 αναφέρονται στοιχεία του 2008 και βρισκόμαστε στο 2010. Ε, θα πρέπει λοιπόν ε, αυτό συμβαίνει συχνά διότι από τη μέρα που λαμβάνουμε μια αναφορά μέχρι τη στιγμή που εξετάζεται περνάει χρόνος αλλά μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για θέματα υγείας να έχουμε λοιπόν πιο φρέσκα στοιχεία τα οποία θα είναι και πιο καθησυχαστικά. Η Ισπανία γνωρίζω πως ε, κατέβαλε ιδιαίτερες προσπάθειες και κάθε φορά έχουμε δεδομένα τα οποία αποκλίνουν. Θα πρέπει λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να λάβουμε νέα στοιχεία για να μπορέσουμε να αποφανθούμε αργότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο υπεύθυνο της ε, Κομισιόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ σε ό,τι φορά την πρώτη παρέμβαση να πω πως συμφωνώ αναφορικά με την ε, ηχορύπανση δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω διότι ακόμα αξιολογούμε τώρα σε φορά την ε, ρύπανση του αέρα επειδή ήμουν σύντομο στην παρουσίασή μου ναι σίγουρα υπήρξε με βελτίωση Κιχών αναφερόμαστε στο 2008 διότι έχουμε τα επίσημα στοιχεία από τη χώρα μέλος μόνο για εκείνη χρονιά. Τα στοιχεία του 2009 θα τα λάβουμε στα τέλη Σεπτεμβρίου εστώτος έτος ε, ίσως ως σχόλιο στην τελευταία παρέμβαση. Πιστεύουμε πως ε, πληροφορίες ε, που θα φτάνουν πιο έγκαιρα θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και για τις εργασίες μας αλλά και για τις ε, σχέσεις και ανταλλαγές με τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν ε, στις, ζητάμε να μας υποβάλλονται εγκαίρως στοιχεία, κάτι το οποίο θα αποβεί προς όφελος όλων μας. Ευχαριστώ. Διατηρούμε ανοιχτές αυτές τις δύο αναφορές και θα εξετάσουμε αργότερα ποιε διαδικασίε θα ακολουθήσουν. Περνάμε στην 18-14-59 του 2007. Ούτε στην περίπτωση αυτή είναι παρόντε οι αναφέροντε. Δίνω το λόγο στον, Κομισιόν, εκπρόσωπο τη Κομισιόν, Πίτερ Βάιντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αφορά την ατμοσφαιρική ρήπανση στην Τεριέστη και σχετικά με την αψηφιακή διασυνορική παράκτια περιοχή της Ιταλίας ε, και την ε, διαχείριση των ε, υδάτων. Αφορά λοιπόν την ρήπανση τόσο του αέρα όσο και των υδάτων. Θα ήθελα να σε τρεις οδηγίες που αφορούν αυτή την υπόθεση IPPC και λοιπά. Τώρα σε ό,τι αφορά την διαχείριση, την οδηγία διαχείριση των ε, υδάτων, έχει ξεκινήσει μια προσφυγή με παραβάση κατά της Ιταλίας λόγω μη συμμάρφωσης για την λόγω οδηγία. Οι αναφερόμενοι αναφέρονται στην γεγονό ότι υπάρχει ελληπή διαχείριση των υδάτων. θέλω να αναφερθώ στο σχόλιο του συναδέλφων για το ζήτημα της ε, ατμοσφαιρικής ρήπανσης υπάρχει μια διαδικασία επί παραβάση και για αυτήν την περίπτωση σε ό,τι αφορά την ρήπανση του αέρα, σε ό,τι αφορά την οδηγία IPPC υπάρχει διμερείς δράσεις. Η Κομισιόν ζήτησε πληροφορίες από την Ιταλία αναφορικά με αυτές τις εγκαταστάσεις και η Ιταλία επιβεβαίωσε ότι η εν λόγω εγκατάσταση διαθέτει άδεια σύμφωνα με την οδηγία IPPC και ε, στην περίπτωση αυτή υπάρχει μια διαδικασία παραβάσης κατά της Ιταλίας γενικότερα για την έλλειψη προόδου στο κράτος αλλά επειδή η εγκατάσταση έχει άδεια δεν ε, θα πρέπει να συνεχιστεί. Οι Ιταλικές αρχές ε, πειδέσαν ότι η εγκατάσταση διαθέτει απαραίτητες ε, τα, τις απαραίτητες άδειες ε, και σε ό,τι φορά τη μη συμμόρφωση θεωρήσαμε ότι η εγκατάσταση θα έπρεπε να κλείσει στα 2009. Ότι αυτή η ψυκάμενος έπρεπε να κλείσει. Δεν ε, υπάρχει κανένα συνάδελφο που επιθυμεί να λάβει τον λόγο σχετικά με τις ε, δύο προσφυγές σε παραβάση αλλά και ό,τι φορά την παρακολούθηση που συνεχίζει η Κομισιόν. Περνάω στην ε, υπαριθμό 19 και στην περίπτωση αυτή ο αναφέρον απουσιάζει. Το λόγο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εδώ το ζήτημα έχει καθαρά τοπικό χαρακτήρα. Πρόκειται για την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στην πόλη Σεύλιεβο και τα συναφή προβλήματα για την υγεία των κατοίκων και το περιβάλλον. Η Κομισιόν Φυσικά έξερα στο ζήτημα της, του θορύβου, της συγχωρήπανσης, αλλά αυτή η οδηγία δεν εμπίπτει, αυτός, αυτή οδός δεν εμπίπτει στην οδηγία περί θορύβου, άρα δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα περί αυτού. Τώρα σε ό,τι φορά την ποιότητα του αέρα, να παραπέμψω στα αρχικά μου σχόλια για τα AS 10 Τώρα, η ε, περιοχή αυτή εκτίθεται σε υψηλά επίπεδα συγκέντρωση σωματιδίων και ειδικά ΑΣ10 και η Βουλγαρία έχει ζητήσει να της παρασχεθεί περισσότερος χρόνος προκειμένου να βελτιώσει την ε, ποιότητα του αέρα Οι βουλγαρικές αρχές δεν κατόρθωσαν να μας πείσουν ότι το στόχο θα τον πετύχουν μέχρι το 2011 όπως είχαν πει. Και γι' αυτό η Επιτροπή θεωρεί ότι θα προβεί στην επιβολή αυτών των ε, οδηγιών όπως έχει κάνει και σε άλλες περιπτώσεις. Ε, νομίζω ότι και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να παραμείνει σε εκκρεμότητα η αναφορά. Περνάμε στην επόμενη, υπερθμονή 20, 553-2007, να ξαναδώσω το λόγο στον Αντρέ Κόμπε. Ευχαριστώ δεν πρόκειται περί τοπικού προβλήματος, αλλά είναι ένα θέμα που αφορά τη Βαρσοβία και κίνηση των πολιτών της Βαρσοβίας κατά της, των σωματιδίων και διοξιδίου του αζότου. Και εδώ θα παραπέμψω στην αρχική μου γενική δήλωση. Οι οριακές τιμές στην Βαρσοβία για τα αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ10 ε, έχουν ξεπεραστεί και τα μέτρα για το διοξείδιο του αζότου θα τεθούν σε ισχύ φέτος, ή σε ισχύ φέτος και δεν ξέρουμε αν έχει σημειωθεί υπέρβαση μέχρι το Σεπτέμβριο 2011. Όσον αφορά τα σωματίδια ΑΣ10, οι πολωνικές αρχές κοινοποίησαν το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πρόγραμμα για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στη Βαρσοβία. Θεωρεί όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η κοινοποίηση δεν είναι επαρκής και προβάλλουμε αντίρρηση όσον αφορά τις παραβιάζονται οι αρχέ τη οδηγία. Δεν ξέρουμε αν οι μετρήσει ήταν επαρκείς πριν το 2005, κατά πόσο οι εξωτερικέ συνθήκε πληρούνται, όπω οι αρνητικέ κλιματολογικέ συνθήκε και τρίτον, κατά πόσο τα μέτρα είναι επαρκή ούτω ώστε να επιτεθεί συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία του 2011. Βάσει αυτή τη αποφάσεω προχωράει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με διαδικασία επιβολή τη νομοθεσία, κάτι που ξεκίνησε και πριν ληφθεί η απόφαση όσον αφορά ε, το θέμα της Βαρσοβίας διότι οι πολωνικές αρχές ε, δεν μας είχαν ε, κοινοποίησει γενικά τα προβλήματα υπέρβαση που είχαν στη χώρα. Ο κ. Ποσινάρου έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μία και μοναδική πτυχή που κατά την άποψή μου είναι πολύ σχετική για τις χώρες αυτές που μπήκαν πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν η οδηγία είναι καλή και ωραία, η διαδικασία της εκτελέσεως της όχι μόνο στην Πολωνία και όχι μόνο σε άλλες χώρες, σε άλλες περιοχές όπως Σερβιεύο, αλλά και αλλού υπάρχει πρόβλημα, όπως και στη Ρουμανία. Πρώτα με την εφαρμογή των ευρωπαϊκών προδιαγραφών και κανονισμών και την αξιοπιστία των διαδικασιών κοινοποίησεως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό μάλιστα όταν υποβάλλεται κάποια αναφορά ή εμφανίζεται κάποια είδη στις εφημερίδες. Το πώς οι κυβερνήσεις και οι αρχές εφαρμόζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες είναι κάτι που παραμένει πάρα πολύ ε, αδύναμο στοιχείο. Και γι' αυτό οι Ευρωπαίοι πολίτες ανησυχούν τόσο πολύ. Όπως με τη βιοπικιλότητα. Ξέρω πολύ καλά ότι στη Ρουμανία και σε πολλά μέρη η εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων ε, είναι πολύ κακή. Και στο τέλος οι Ευρωπαίοι πολίτες κατηγορούν και σωστά με επιχειρήματα και χωρίς επιχειρήματα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ συνάδελφε Μποσινάρου, αν δεν θέλει να πάρει άλλο το λόγο, αφήνουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά. Συνεχίζουμε με την αναφορά 21 τη 1066 του 2008 στον κύριο Πρόιζη δίνουμε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σε αυτή την υπόθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ότι το Open University, το ανοιχτό πανεπιστήμιο, που χορηγεί μαθήματα εξ αποστάσεως εφαρμόζει ανισότητα όσον αφορά τις εγγραφές πιο ψηλές τιμές ε, απαιτεί από αυτούς που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί της Υπήρου της Ευρωπαϊκής και πιο μικρή τιμή για όσους είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο και πιο ψηλή τιμή λίγο για αυτούς που μένουν στην Ιρλανδία. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέδειξε ότι αυτό εξηγείται εν μέρη από τότε η κυβερνητική χρηματοδότηση της ανώτατης παιδείας στο Ηνωμένο Βασίλειο βασιζόταν σε κριτήρια που αφορούσαν τον αριθμό των σπουδαστών, των γεγραμμένων και που διαμένουν στα πανεπιστήμια. Όμως αυτό γίνεται για όλα τα Βρετανικά πανεπιστήμια που υποδέχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο τους σπουδαστές που θέλουν να παρακολουθεί τα μαθήματα. Όμως το Open University είναι ένα ίδρυμα που κάνει διδασκαλία εξ αποστάσεως. Οπότε αυτοί που δεν διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν αποτελούν τμήμα της, των κριτηρίων της δημόσιας χρηματοδότησης και το Open University ε, ζητά περισσότερα χρήματα για την εγγραφή. Το δίκαιο της ε, ενώσεως είναι το άρθρο 20 και το άρθρο 18. Το άρθρο 20 που καθορίζει την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και δίνει σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη το δικαίωμα ε, να μην είναι αντικείμενο διακρίσεως λόγω επικότητας όσον αφορά τον τομέα που εφαρμόζει τη ησυχία. Το άρθρο 65 του 2 της συνθήκης διευκρινίζει ότι η δράση της ενώσεως θέλει να ενθαρρύνει την εξαποστάσεως διδασκαλία. Και αν διαβάσουμε τα τρία άρθρα μαζί, μα οδηγεί στο συμπέρασμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η άνηση αντιμετώπιση που διαπιστώνεται αποτελεί έμεση διάκριση λόγω ε, Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά διαδικασία παράβασης και γίνονται ε, επαφέ μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι δυνατόν να δώσουν περισσότερε πληροφορίε επί του παρόντο, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορέσει να συμμορφωθεί ε, με το κοινοτικό δίκαιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι σε θέση να δώσει στο δεύτερο εξάμεινο ενεστώτο έτου περισσότερε ε, πληροφορίε. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιο να πάρει το λόγο. Ναι, διότι διαπιστώνω κάτι. Πρόκειται περί αναφοράς του 2008 και είμαστε σήμερα τρίτη ε, του 2010. Μία τρίτη του 2010. Και διερωτώ με, πόσος χρόνος απαιτείται για να χειριστούμε μια τέτοια κατάσταση που αναφέρθηκε ότι είναι σαφής, ε, αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι σαφής η κατάσταση αποδεικνύεται ότι πρόκειται περί παραβάσεως και το διαπιστώνει αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2008, 2009, 2010. Πού είναι η αποτελεσματικότητα και πώς υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών μας είναι ένα ερωτηματικό. Ελπίζω ότι τελικά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δρά πιο αποτελεσματικά. Είναι ανάγκη αυτό πιο πραγματιστικά. Είναι κάτι απαραίτητο. Διαφορετικά, η ίδια κατάσταση θα ισχύει και σε όσες άλλες περιπτώσεις. Έχουμε πολλές εξηγήσει, όμως οι εξηγήσει δεν είναι πάντα η απάντηση που περιμένουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και που χρειάζονται. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν κατάλαβα σωστά αν απευθύνατε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αίτημά σας, την έκκλησή σας και εγώ συμφωνώ, εσείς υποστηρίζω σε αυτή την έκκλησή σας. Τέλεια. Συμφωνώ με την έκκληση του συναδέλφου Μποσινάρου. Αφήνουμε ανοιχτή την αναφορά. Εν αναμονή ε, των αποτελεσμάτων τη δικασία παράβαση. Τελευταίο σημείο τη σημερινής διάταξη, η αναφορά 683 του 2009. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Λαβρέντζου τον κύριο Λαβρέντσο. Euh, Με ακούτε τώρα. Λοιπόν, αυτή η αναφορά αφορά Ιταλούς φοιτητέ και αφορά στον αριθμό των ε, μονάδων που έχουν συλλέξει σε ό,τι αφορά την ισοδυναμία, ισοδυναμία των πτυχίων Ιταλικών Πανεπιστημίων σε ορισμένα κράτη-μέλη και θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα για τη μεταφορά ε, πόντων ή e CTS. Σύμφωνα λοιπόν με τους αναφερόντες, οι μελέτες τους στην Ιταλία θα δώσουν 300 μονάδες ενώ όταν πήγαν στη Σουηδία, στη Δανία και στο Ενωμένο Βασίλειο έλαβαν από 180 έως 240 μονάδες. Κάτι το οποίο θεωρούν ότι δεν είναι αρκετό. Ξέρετε πως ε, υπήρξε μεγάλη πρόοδος ε, σε αυτά τα ζητήματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε θέματα εκπαίδευσης. Υπήρχαν εποχές όπου ήταν δύσκολο να, ακούσουμε, να προβούμε σε μια διαδικασία ε, επί παραβάση. δεν μπορούμε να το πράξουμε διότι δεν υπάρχουν υποχρεωτικοί κανόνες αλλά αυτό το οποίο λέμε είναι πως οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε ζητήματα ισοτιμίας και αναγνώρισης από τα πανεπιστημιακά δρήματα ή από άλλες αρχές θα πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να υπάρχει δυνατότητα ε, προσφυγής ε, τώρα. Υπάρχει υψηλό αριθμό πανεπιστημίων στην Ευρώπη και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο υπολογισμό να μην γίνεται πάντα εύκολα και να μην ακριβή. Η Κομισιόν λοιπόν επιθυμεί να υπάρξει διαφάνεια, υπήρξε προς ζήτημα, αλλά δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε πως ε, σε κάθε περίπτωση ένας φοιτητή ο οποίο μεταβαίνει στη Σουηδία να την χάνει ενό υπολογισμού των μονάδων του με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται σε άλλο κράτος μέλους. Έχουμε εδώ το, την απάντηση που τον στείλαμε στους 55 έχει στείλω επίσης ε, και έναν οδηγό είναι οδηγό χρήστη όπου αναφέρονται όλα τα πράγματα με σαφή τρόπο. Αναφερθήκαμε στις σελίδες ε, που τους αφορούν ιδιαίτερα, τους, τους 55 φοιτητές. Αυτά μπόρεσε να κάνει η Κομισιόν μέχρι τώρα για το ζήτημα. Επιθυμεί κάποιος συνάδελφος να λάβει το λόγο. Γκρούνε. Θα ήθελα να πω ότι είναι ουσιώδες ε, να απαντήσουμε στους ε, Ευρωπαίους πολίτες. Οικοδομούν την Ευρώπη για λογαριασμό τους. Η Ευρώπη για μένα είναι ένας μεγάλος χώρος ε, ελευθερίας και όταν παρατηρούμε τις δυσκολίες που υπάρχουν στην αναγνώριση πτυχίων, διότι συχνά λαμβάνουμε αναφορές ή όπως στην περίπτωση αυτή για τις ισοδυναμίες ε, και για τις μονάδες ε, που εξαρτάται από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο κλπ. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει λοιπόν ε, να δραστηριοποιηθούμε προκειμένου να υπάρξει πρόοδος στα κράτη-μέλη και να ανταποκριθούμε στα αιτήματα και τις προσδοκίες των νέων μας. Είναι ανάγκη Πρόεδρος, ε, συμφωνώ με τις παρατηρήσεις της ε, συνάδελφου, γκρούνι Γκρούνη και θα πρέπει κάπως ε, να προβληματιστούμε σχετικά με αναφορές που έχουν παρόμοιες παρόμοιο ή παρεφερές αντικείμενο. Εδώ μιλάμε για τις μονάδες, σε άλλες αναφορές μιλάμε για τις ισοδυναμίες, τις ισοτιμίες, αναγνώριση κλπ. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που αφορά υπηρεσίες. Εμεί θέλουμε να εγγυηθούμε την ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών και θεωρώ ότι μπορούμε να, μπορεί η Κομισιόν να κάνει περισσότερα πράγματα από ότι να αποστείλει ένα, μια ιστοσελίδα στους φοιτητέ που μπορεί να τους ενημερώσει για το πρόβλημά τους. Λοιπόν, ξεκινώντας ε, από αυτή την αναφορά θα ήθελα να προτείνω να την διατηρήσουμε ανοιχτή για να το ξανασκεφτούμε και να δούμε πού μπορούμε να οδηγηθούμε. Εκτός αν κρίνεται ότι θέλουμε, μπορούμε να την κλείσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δεσμευτούμε να εξετάσουμε το ζήτημα και να προβληματιστούμε περαιτέρω. Να κλείσουμε λοιπόν την αναφορά και να εξετάσουμε... Όχι, όχι. Ανοιχτή λοιπόν θα παραμείνει η αναφορά και θα αξιολογήσουμε με τους συντονιστές ε, ποιος ήταν ο καλύτερος τρόπος για να εμβαθύνουμε περαιτέρω το ζήτημα. Ε, Ξαντλήσαμε σε χρόνο ρεκόρ την μέσα διάταξη. Ως εκ τούτου μπορούμε να κηρύξουμε το πέρας ε, της συνεδριάσεως της Επιτροπής μας. Α, per quanto riguarda... Σε ό,τι αφορά το δεύτερο τμήμα της ημερησίας διατάξεως υπάρχει αίτημα της συναδέλφου Όκεν για το σημείο 32. Είναι το μοναδικό θέμα λοιπόν που βγαίνει από το τμήμα Β.